Ωραία λοιπόν. Για ναι, να δούμε σιγά σιγά να ανασύντασόμεθα. Um, so... Δεν θα ψηφίσουμε ακόμα, οπότε τι η αναταραχή. Okay. Uh, right, we're on to point... Ερχόμαστε στο σημείο 11 τώρα. που είναι η έκθεση του Πάμπλο ποινική προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη θα παρουσιάσει την έκθεσή του ε, από πλευράς Προεδρείου. Ε, ευχαριστώ πολύ Σάρων. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ε, η εναρμόνιση του συστήματος, ο εξυγχρονισμός και η βελτίωση για την ποινική προστασία ε, από την παραχάραξη όχι μόνο του ευρώ και των άλλων νομισμάτων. Είναι κανονισμός 1338 ε, κάθετος 2001. Γενικά υποστηρίζουμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία και ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με την εναρμόνιση αλλά και τις κυρώσεις και σε καιρούς κρίσεων προφανώς αυτό είναι όθηση για την καταπολέμηση της απάτης και όσο πιο συντονισμένες και ε, ενωμένες είναι κινήσεις αυτές τόσο το καλύτερο. Ο συντονισμός ε, και η συνεργασία είναι πάρα πολύ εύλογος εδώ γιατί το ευρώ έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, για την οικονομική και νομισματική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας στο ευρώ. Και γι' αυτό θα πρέπει να εγγυηθούμε την καλή προστασία του νομίσματος μας, των πολιτών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση τι φιλοδοξία έχει. Όλα τα κράτη-μέλη να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις και τους ίδιους όρους μέσω συνεργασίας στόχος είναι να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια ε, με ευθυγράμμιση ε, σε άλλες εκθέσεις Επιτροπής ΕΚΟΝ, όπως να δημοσιεύονται οι καταδίκες για να έχουν και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Επίσης να υπάρχει αναλογικότητα των ποινών και των κυρώσεων ε, με βάση την αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσης θέλαμε να έχουμε ενία, μάλλον συνεπή εφαρμογή, ευρεία, ε, παραχάραξη όχι μόνο των χαρτονομισμάτων αλλά και των κερμάτων ε, και όχι μόνο του ευρώ αλλά και άλλων νομισμάτων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αδικήματα ε, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την νομοθεσία, να την αυστηροποιήσουμε, αλλά και ε, να διευκολύνουμε την ανταλλαγή προφοριών και το πιο στενό ε, συντονισμό των διοκτικών αρχών για να υπάρχει και πιο αποτελεσματική δράση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έκαναν τροπολογίες, την Ελίζα Φερέιρα, τον Ashley Fox, τη Σιλβί Γκουλά, τον Ζαν Οντί και ακολουθεί μακρύς κατάλογος συναδέλφων. Ε, είχαμε επίσης συναντήσεις με όλους ε, τους συντάκτες ή ε, τους εκπροσώπους τους για να συμφωνήσουμε. Και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ελίσσα. ευχαριστώ Σάρον. Δεν έχω και πάρα πολλά να προσθέσω σε σχέση με αυτά που μας είπε ο συνάδελφος Παύλο. Ήθελα μόνο να τονίσω ότι αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντική στο μέτρο που ενισχύει το σύστημα κυρώσεων σε σχέση με την ε, κινδυλία των νομισμάτων και την παραχάραξη των χαρτονομισμάτων συμπεριλαμβανομένου και του ευρώ και άρα έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα, λίαν αποτρεπτικό χαρακτήρα και εξαιρετικά επίκαιρο και ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή, ήταν εξαιρετική η δουλειά που έκανε. Και πιστεύω ότι οι τροπολογίες που καταθέτει και αυτές που θα καταθέσουμε και εμείς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είναι τέτοια φύσης ώστε να βελτιώσουν την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ήθελα να τονίσω και δύο πτυχές του ζητήματος, πέρα από αυτό που μας είπε ο εισηγητής. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δημοσιοποίηση των καταδικαστικών αποφάσεων, γιατί έτσι ενισχύεται ο αποτρεπτικός χαρακτήρας ε, των μέτρων και προβάλλονται αυτά τα μέτρα. Ε, επίσης, ε, για την ποινικοποίηση της μη ολοκληρωμένης παραχάραξης και της παραχάραξης άλλων νομισμάτων θα καλύπτονται έτσι καλύτερα. Αυτά και άλλα θα συμπεριλαμβάνονται στις τροπολογίες ε, που θα εξετάσουμε σε συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδης. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι βελτιώνουν όλες αυτές τις τροπολογίες το περιεχόμενο της αρχικής πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δημόσια λοιπόν ε, ε, εκφράζω την υποστήριξή μας για την συνενετική αυτή θέση. Και όπως είπαμε και στη τελευταία σύσκεψη των ε, σκιωδών ε, θα καταθέσουμε και άλλες τροπολογίες αλλά πραγματικά πιστεύω ότι βελτιώνουμε την αρχή πρόταση Επιτροπής και επιδιώκουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους ε, προδιαγραφέτες στόχους. Ευχαριστούμε. Ε, ε, από τους φιλελεύθερους έχουμε κάποιον. Πράσινη. Λάμπερτς. Ο Ρούι έλεγε τα βάρες ότι ναι, ναι, δεν είμαι ο Ρούι. Αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να μιλήσω. Βουλευτής είμαι. Θα μιλήσω λοιπόν. Ε, ούτε να ευχαριστήσω ούτε να συγχαρώ τον εισηγητή δεν θέλω διότι είτε θα πρέπει να τον επικρίνω για έλλειψη θάρρους, δεν έκανε καμία αμφιλεγόμενη πρόταση ή θα πρέπει να τον ευχαριστήσω διότι συμπαρατάθηκε με τους πράσινους. Ή αλλιώ δεν είναι αμφιλεγόμενο το ζήτημα, οπότε τι, με τι ασχολούμαστε. Δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα και σταματά εδώ. Ολέ, κάτι σου ήρθε τώρα, θέλεις και εσύ να προσθέσεις κάτι. Δεν θα έπρεπε ίσως γιατί εμείς έχουμε άλλο νόμισμα, αλλά τέλος πάντων. Στην Επιτροπή για την Οργανωμένη Εγκληματικότητα ΚΡΙΜ μιλήσαμε για 500 χαρτονομίσματα. Α, συγγνώμη, το, ε, το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Ε, άρα πρέπει να καλυφθούν και οι παράνομες ε, δραστηριότητες. Ωραία, λέει η Πρόεδρος. Τότε να επιστρέψουμε στον Άσλεϊ στους ε, επίσημους δηλαδή σκιώδεις. Απογοητεύτηκα λίγο γιατί δεν πέρασε καμία από τις τροπολογίες μου. είναι σημαντικό να ε, προστατεύσουμε όχι μόνο το ευρώ αλλά και τα υπόλοιπα νομίσματα από τις απάτες. Όμως ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η αρχή της επικουρικότητας. Και νομίζω ότι παραβιάζεται αυτή η αρχή, διότι εισάγονται ελάχιστες ποινές. Ε, οι ελάχιστες ποινές, το ποινικό δίκαιο γενικότερα, καλύτερα να επαφίεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και γι' αυτό εμείς δεν πρόκειται να υποστηρίξουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Άλλος. Κάποιος από την Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Είναι πολύ πιστική και επικοδομητική η έκθεση. Μπορούμε να υποστηρίξουμε μεγάλο μέρος των Κυρίως ε, τη θέση του εισηγητή Κοντ και των σκιωδών για τις ελάχιστες κυρώσεις. Εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος αυτό το στοιχείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ελάχιστα ε, πρότυπα για τις ανώτατες ποινές, τις ανώτατες κυρώσεις είναι μια ιδέα που υποστηρίζει εμπολής ο εισηγητής και ε, θέλουμε να καλύψουμε και τα ε, παραγωγικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παραχάραξη. Θέλουμε επίσης να παραμείνει η μνήα στη Σύμβαση της ε, Γενέβης σε αυτό το νομοθέτημα, διότι έχει μεγάλη σημασία για την εφαρμοσιμότητα της αρχής της μη διακριτικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα. Για αυτή την πρόταση και όχι μόνο για αυτή, βασιζόμαστε στη Σύμβαση της Γενέβης και σε αυτή την αρχή. Μας ικανοποιεί λοιπόν και η έκθεση και οι τροπολογίες. Ε, πολύ σύντομα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, λέει ο κύριος Σάλμπα. Ευχαριστώ και το Φίλιπ Λάμπερτς. Δεν ξέρω αυτό είναι υποστήριξη από πλευρά πρασίνων 100% υποστηρίζετε το ΕΛΚ μήπω και μπείτε στη γερμανική κυβέρνηση. Λέω τώρα. Πάντως με χαρά άκουσα τα σχόλιά σας. Ε, για το χαρτονόμισμα των 500 ε, ευρώ ε, θα το σημειώσουμε. Και αυτό που ζήτησε η Σιλβή και για τα 200 ευρώ. Συμφωνώ με αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό αυτό για την προστασία ε, του ευρώ και σε σχέση με το όσο είπε ο Άσλη, ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες. Ε, θα βρούμε μια συμβαστική πρόταση για ε, τις κατώτατες ποινές ή τα πρόστιμα. Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε, θα προσπαθήσουμε ε, να τα βρούμε και στα υπόλοιπα ζητήματα που εκκρεμούν. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας και με χαρά συνεργαστήκαμε με όλους εσάς. Very much. Ε, ευχαριστώ πολύ. Στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε στις 24 το μηνός που είναι σήμερα εντός ολίγου, εντός ολίγων λεπτών. Στην... Στις 3 Οκτωβρίου ψηφίζει ε, ε, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και αργότερα στην Ολομέλεια. Τελειώσαμε ακριβώς την ώρα μας και πάμε μέσω στην ψηφοφορία. Αν είναι όλα έτοιμα, έχετε όλες τις κάρτες σας. Okay, if you've got your cards, can you plug them in? Ωραία, λοιπόν, έχετε τις κάρτες σας, τις βάζετε στην σχέση που πρέπει. Ας κάνουμε μια δοκιμή, πατήστε το ε, κουμπί να ψηφίζετε. Δοκιμή τώρα. Ε, η πρόεδρος Α, τώρα μόλι κατάφερα να κάνει το δικό μου σύστημα να λειτουργήσει. Ωραία, ποιος ε, του λείπει η κάρτα του, ποιο θα έχει ξεχάσει την κάρτα του, κύριο. Οντομάν, Σφέν. να φροντίσετε να ψηφίζετε αντίθετο ένα από τον άλλο, εσεί οι δύο που δεν έχετε κάρτα. Τώρα απ' την άλλη, αν ψάχνετε να φτιάξετε συμμαχίε. Μπορεί τα αποτελέσματα τη ψηφοφορία να είναι ενδιαφέροντα. Εσεί το ξεκινήσατε αυτό, ε, το αστείο. Σα είδα που μιλούσατε πριν. Όλο φιλοφρονήσεις είμαστε. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. Ε, τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Ε, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία συμβιβαστική α υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν εγκρίνεται, α πούμε. 59 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 Οπ, ε, με συγχωρείτε ε, εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπέρκατα, 70 υπέρ, γκρίνεται, 71 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική E υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. F υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ ε, Θεόδωρος. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για τις 8 και 76 θέλω να σφιστήσω τη προσοχή σας στο γεγονό ότι είναι ίδιες. Ε, επιδιώξαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης να διαγράψουμε την αναφορά στις κατεξουσιοδότηση πράξεις που δίναμε αυτή τη δυνατότητα στην Επιτροπή. Λάβαμε τη γνωμοδότηση όμως της νομικής υπηρεσίας και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανέλθουμε Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που από νομική απόψεως πρέπει να είναι πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Άρα εδώ η θέση μα είναι κατά. Θα μπορούσατε να την είχατε αποσύρει, λέει η πρόεδρος. Τέλος πάντων. Ωραία, άρα ο εισηγητή ζητάει να καταψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτονται λοιπόν. 77 υπέρ. Κατά. Με μπερδέψατε. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Έναρξη έναξη Συν ένα μείον ένα. Από εκείνους που δεν έχουμε κάρτες. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει σημασία, ε, συμμαχία μεταξύ των πρασίνων και του ΕΛΚ. Δεν χρειάζεται να ψηφίσω εγώ λοιπόν, λέει η πρόεδρος. Πρόεδρος υπήρχε συν ένα, μείον ένα. Δεν υπάρχει συμμαχία μεταξύ τους, σου λέω. Άρα απορρίπτεται. Υπέρ 21, λοιπόν 9 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε. Λοιπόν, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 11. Λήξη ψηφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική I, J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική K, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. L, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. M, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται εγκρίνεται εν υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται Τρόλη 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά, κατά αποχές απορρίπτεται η 30 συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τεσ. Και πάμε στην Q. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στην R, συμβαστική R, υπέρ, κατά τα αποχές εγκρίνεται. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα ηλεκτρονικό, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία για, για το σύνολο της πρότασης. Για το, να εκθέσει όπως τροποποιήθηκε. Ένα ψηφοφορίας. Λήξη. 42 υπέρ και μία αποχή. Συγχωρείτε, συν δύο ε, συνάδελφοι που δεν είχαν την κάρτα τους, άρα 44 υπέρ, καμία, κανένας κατά, μία αποχή. Και τώρα επί του ψηφίσματος, πάλι ηλεκτρονικά, έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Και είναι το ίδιο αποτέλεσμα. 44 υπέρ, κανένας κατά, μια αποχή. Συγχαρητήρια. Όχι, τώρα πρέπει να ψηφίσουμε για την εντολή διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό 70. Ο εισηγητής θέλετε να μιλήσετε. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιώδες και όλους τους ε, συναδέλφους για τη συνεργασία. Ήταν ένα θέμα λεπτό και δέστητο. Ελπιστώ ότι στον τριμερή διάλογο θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη θέση μας. Και προτείνω να πάμε στον τριμερή διάλογο και όχι στην Ολομέλεια. Πρόεδρος, ωραία. Άρα η πρόταση του εισηγητή είναι να ξεκινήσουμε ε, πρώτη ανάγνωση για ε, στόχο να καταλήξουμε σε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης με εντολή την έκθεση που μόλις υπερψηφίσαμε και σύνθεση της ε, διαπραγματευτικής ομάδας, συνήθις, δηλαδή πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ο εισηγητής και οι σκιώδης. Μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά από αυτού. Αν ψηφίσετε υπέρ σημαίνει ότι συμφωνείτε, δηλαδή να ξεκινήσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ε, ψήφισαν όλοι 41 υπέρ, 40... μάλλον, συν του δύο συναδέλφου που δεν είχαν κάρτα. 43 υπέρ λοιπόν, 3 κατά, καμία αποχή όσο πάει και γίνεται πιο περίπλοκο αυτό το πράγμα με την ψηφοφορία, λέει η πρόεδρο. Πάμε στο επόμενο σημείο της τη διάταξη, σημείο 13. Ε, προστασία του ευρώ και άλλων ε, νομισμάτων, δηλαδή η έκθεση που μόλις συζητήσαμε από την πλαστογραφία. Όλοι είναι έτοιμοι. Ωραία. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Όχι, με, με συγχωρείτε λέει πρόεδρος, 14 καταπίπτει. 6 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, 8 λοιπόν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 έχει αποσυρθεί 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 έχει αποσυρθεί και ψηφίζουμε για την 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε τη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι λοιπόν 41 υπέρ 4, 4 κατά μία αποχή. Ωραία. We're a bit early for Mr. Taylor's report. Does that matter? Hmm?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 Okay, um, Mr. Pitella, who is the... Κύριε είστε εισηγητής για την ετήσια έκθεση ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά δεν έχει καταστάσει ο κύριος Πιτέλα, γιατί προεδρεύει σε μια συνδιαλλαγή και εμείς ε, τελειώσαμε νωρίτερα. Πεντάλεπτη διακοπή, για να ξέρετε τι συμβαίνει, περιμένετε άδικα. ο σκοπός μας είναι να τελειώσουμε και νωρίτερα, οπότε ας μην το παρακάνουμε με το διάλειμμα να είναι σύντομο. Okay. Ήρθε ο κύριος Πιτέλα. Δεν άργησε, εμείς τελειώσαμε νωρίτερα. Ας ε, χρησιμοποιήσουμε όμως αυτό το χρόνο. Παρακαλώ να κάνετε περισσότερη ησυχία όσοι κάνετε αυτά τα πηγαδάκια εκεί πίσω. Πρόκειται για μία έκθεση για την ΕΚΤ, για τους ετήσιους λογαριασμούς του 2012, αλλά ως συνήθως θα θέλετε να πείτε και κάποια πράγματα για το 2013, συνήθως δεν συγκρατούμαστε και δεν αυτοπεριοριζόμαστε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να μας παρουσιάσει ε, την έκθεσή του. Τζάνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για την ε, υπομονή τους, ε, αλλά γινόταν η συνδιαλλαγή και για τον προϋπολογισμό και είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθώ σε όλα ταυτόχρονα. Θα ήθελα να δηλώσω ευγνώμων προς όλους τους συναδέλφους όλων των πολιτικών ομάδων για 247 τροπολογίες που κατέθεσαν. Ε, μετά από μια πρώτη ανάλυση των τροπολογιών, έχω την εντύπωση ότι έξι είναι τα κεντρικά ζητήματα από τις πλευράς ε, του ΕΛΚ, των σοσιαλιστών και των φιλελευθέρων. Να γνωρίζετε ο θετικός ρόλος ε, της ΕΚΤ κυρίως μέσα από το πρόγραμμα για τη σταθεροποίηση τη της Ευρωζώνης. Επίσης, Ζητείτε μεγαλύτερη διαφάνεια και ανάληψη περισσότερων ευθυνών από το ΕΚΤΕ και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση, στην νέα αρχιτεκτονική δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνει νέα, νέες αρμοδιότητες, νέα καθήκοντα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άρα θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Φέλτσα για την τροπολογία της διότι μας ε, ζητάει ε, ε, πρακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, παραδείγματος χάρη της ΕΚΤ. Στη συνέχεια, σε άλλες τροπολογίες βλέπουμε ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες ε, στην ε, πραγματική οικονομία ω προς τις επιχειρήσεις. Ε, βλέπετε αυτέ τι πληροφορίε στι διαφορέ τροπολογίες. Η υιοθέτηση προγραμμάτων αντιστοίχων με το Μνημόνιο της Ελλάδας, πρόταση του κυρίου Τόρβαλς παραδείγματος χάρη, εκεί ζητείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ασχοληθεί και με τις bank securities, έτσι αναφέρει η τροπολογία. Υπάρχουν πολιτικές λιτότητες ιδιαίτερα αυστηρίες, ε, ε, οι σοσιαλιστές ε, και οι γκούε θεωρούν αντίθετα με τις υπόλοιπες τρεις πολιτικές ομάδες ότι πρέπει να προβούμε σε αναθεώρηση του ιστορικού ε, καταστατικού της ΕΚΤ ούτως ώστε ο βασικός στόχος και μοναδικός στόχος να είναι η σταθερότητα των τιμών. Ε, ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ε, βιώνουμε αυτή τη στιγμή ριζική ε, μεταρρύθμιση του παγκοσμίου νομισματικού συστήματος. Ε, η τροπολογία της ε, κυρίας Γκάλ ε, για αυτό το λόγο είναι εξαιρετική βάση συζήτησης. Θα ήθελα δεν να σταματήσω εδώ και να συζητήσουμε λεπτομερέστερα την επόμενη Πέμπτη με τους σκιώδες άλλες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ας ακούσουμε τώρα τους σκιώδες από το ΕΛΚ. Η κυρία Γκάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή για τη δουλειά όλη αυτή που έκανε. Έχουν γίνει πάρα πολλές τροπολογίες που μπορούν να ταξινομηθούν ε, σε κατηγορίες όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν, δεν είναι τίποτα καινούριο. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να ε, δημιουργήσουμε ε, μια ε, προστιθέμενη αξία. Επιτρέψτε μου μερικά σχόλια, όχι μόνο για τις τροπολογίες γενικά. Ποια ήταν η αφετηρία μας. Όπως και πέρυσι, η ετήσια έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας και που τονίζουμε και επιμένουμε να περιγράφεται σωστά ε, και με σαφήνεια η λειτουργία και τα καθήκοντα της τράπεζας. Η συνθήκη τα λέει αυτά και θα πρέπει να τα τηρούμε στα διάφορα κράτη-μέλη. Κυριαρχεί το θέμα της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ε, τη δημιουργία νέων δομών δανειοδότησης, αλλά αυτό δεν είναι βασική ενασχόληση, ούτε το πρώτο καθήκον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μπορεί να είναι ευσεβής πόθη ορισμένων, αλλά δεν είναι η δική μας δουλειά αυτή. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έπαιζε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν επενέβη στην περίπτωση των OMT ε, και φρόντισε να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως όφιλε. Εξασφάλισε τη σταθερότητα του ευρώ. Ε, μπορεί να διαπιστωθεί αυτό και να σημειωθεί ως παρατήρηση χωρίς ε, περαιτέρω ανάλυση. Τον Ιούνιο επίσης προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων. Συμφωνώ και με αυτό. Αλλά συμφωνώ και με τους συναδέλφους που λέγουν ότι όταν τα επιτόκια παραμένουν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα πολύ χαμηλά, στο αυτό είναι αρνητικό. Σε ό,τι αφορά την αιρεσιμότητα, εγώ θεωρώ ότι η πραγματική οικονομία δεν χρειάζεται όρους και προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα θα μπορεί ε, από μόνη της να ανακάμπτει κανονικά. Αυτό δεν είναι ο ρόλος της. Και εκτός αυτού θα πρέπει να προχωρήσουμε σε νέα μέτρα ε, για να ε, επιτύχει αυτή η ε, μεταβατική περίοδος και να μειωθούν τα πολύ ψηλά επιτόκια με τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να δανειζόμαστε ορισμένοι. Ε, ε, στην πραγματική οικονομία δεν γεννήθηκαν τα περισσότερα προβλήματα λόγω έλλειψης δανειοδότησης. Είναι ένα τμήμα του προβλήματος. Και σε ό,τι φορά το πρόγραμμα χρεογράφων είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να τονίσω κατά τα άλλα ότι σε σχέση με τα προβλήματα των διαφόρων κυβερνήσεων δεν είναι η λύση όλων μας των προβλημάτων γιατί δεν είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, εξηγένει τους ε, προϋπολογισμούς των κρατών μελών ή να αυξάνει το έπτους. Χαίρομαι γενικά για τα μέτρα αυτά και για τον τρόπο που εφαρμόζονται χωρίς και τιμές. Στο προσεχές μέλλον ε, θα πρέπει να συνδέονται πολύ με όρους και προϋποθέσεις και με πολύ αυστηρούς μάλιστα. Συμφωνώ με τους συναδέλφους. που έκαναν προτάσεις για μεγαλύτερες διευκολύνσεις. Και υποστηρίζω την άποψη που λέγει ότι η Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει σιγά σιγά να χαλαρώνει την πίεση όσο χαλαρώνουν και οι εντάσεις στις αγορές. Δεν μπορώ να υποστηρίξω όμως τις τροπολογίες που θέλουν να αυξήσουν το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας για το πληθωρισμό, ανεξάρτητα για ποιο λόγο. Ενδεχομένως για να ξεγειάνουν τους προϋπολογισμούς των κρατών, αλλά για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να έχει μια δημοκρατική διοίκηση, αλλά φαντάζομαι αυτή τη διακυβέρνηση με κάπως διαφορετικό τρόπο από ορισμένες τροπολογίες και πιστεύω προσωπικά ότι η ανεξαρτησία της τράπεζας μπορεί να υλοποιηθεί κατά δεύτερο λόγο. Και δεν είναι η βασική μέρημνα της Κεντρικής Τράπεζας. Κατά τα άλλα υποστηρίζω την πρόταση του εισηγητή να υπάρχει ένας εντατικός νομισματικός διάλογος. Το έχουμε ξαναπεί εδώ επανειλημμένα, όπως και στην Ολομέλεια άλλωστε. Οι νέες εποπτικές ε, αρμοδιότητες ε, στην Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να είναι ξεχωριστές. Μια τελευταία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Στη συνεδρία των σκιωδών θα ε, ε, συνεχίσουμε τη συζήτηση για τις τροπολογίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους οι διάφοροι θεσμοί ή τα θεσμικά όργανα που έχουν να κάνουν με την νομισματική πολιτική. Έχουν γίνει πολλές τροπολογίες. Ως προς το ρόλο του ευρώ ως διεθνές νόμισμα ή το ρόλο των γυναικών ε, στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά αυτά δεν είναι του παρόντος, θα τα πούμε σε άλλη συνεδριάση των σχεδόν. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, LD group, Neil Torvalds. Neil Torvalds, ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή πρώτα απ' όλα για την ε, έκθεσή του. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες για όλες τις τροπολογίες, ε, διότι κάποιες ε, δεν θα συζητηθούν εδώ και κάποιες είναι άσχετες με το αντικείμενο. Δύο-τρεις μόνο θέλω να σχολιάσω. Πρώτα απ' όλα, δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε τώρα να ε, ξεφύγουμε από το πλαίσιο της έκθεσης και να ζητήσουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Διότι στην τροπολογία που έχουμε για την πολιτική και ακαδημαϊκή συζήτηση ε, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να το τονίσουμε αυτό μέσα στην έκθεση. Όχι ότι έχω και κάτι κατά, μπορούμε να το ζητήσουμε, αλλά Σίγουρα εμείς δεν θα υποστηρίξουμε κανένα αίτημα αναθεώρησης συνθήκης σε αυτό το στάδιο, παρότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση και γι' αυτό. Δεύτερον, το θέμα των συλλαγματικών ισοτιμιών και της ε, πολιτικής των ε, ισοτιμιών είναι διακρατικό το ζήτημα ή για να είμαι πιο συγκεκριμένος ε, ζήτημα ε, του, τον, του οικονομικού τομέα της κάθε χώρας. Θυμάστε τη δεκαετία του 70 όταν ε, προσπαθήσαμε να λύσουμε οικονομικά προβλήματα υποτιμώντας σημαίνει τα νομίσματα σε σχέση με τους δε. Ε, και ε, αναθερμάνθηκε όντως η οικονομία αλλά μετά γρήγορα πάγωσε και γίνανε χειρότερα τα πράγματα. Εμείς έτσι ε, προσεγγίζουμε το, το θέμα, ε, υποστηρίζουμε τις τροπολογίες 14-16. Το τρίτο ζήτημα είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία. Όλοι Όλοι υπογραμμίζουμε ότι ε, είναι απαραίτητη ε, η λογοδεσία, αλλά όχι να χρησιμοποιηθεί και ως φίλος εκεί για να καταστεί ε, λιγότερο αμερόληπτη η ΕΚΤ. Το αντίθετο. Χτες ακούσαμε τον κύριο Ντράγκη να μας λέει ότι τελικά κανείς δεν ξέρει ποιος παίρνει την, τελευταία, την τελική απόφαση. Δεν θα μας έβλαπτε λίγη περισσότερη διαφάνεια όταν μιλάμε για το ρόλο τρόικα της, του, ε, της Καλά κάνουμε και το αναφέρουμε στο σχετικό τμήμα της ε, έκθεσης. Ε, νομίζω ότι με τη συζήτηση θα καταφέρουμε τελικά να ρυθμίσουμε τα εκρεμή ζητήματα. Ευχαριστούμε. Η πράσινη Σβέν. Η, η σκιώδης μας, η Εύα Ζολή, δεν μπορεί να έρθει. Θα σας διαβάσω τη δήλωσή της. Σας ευχαριστώ για το σχέδιο έκθεσης που είναι εξαιρετική βάση εργασίας για την ε, τελική έκθεση. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στην εμπλοκή της έκθεσης στην Τρόικα μέσα στο σχέδιο έκθεσης και γι' αυτό ζητάμε ε, αξιολόγηση του μόντους οπεράντη της Τρόικα και της εμπλοκής ε, της έκθεσης σε αυτό το πλαίσιο. Είναι της σημασίας η διευκρίνηση και επαναπροσδιορισμός του πεδίου και των αρμοδιοτήτων και της δημοκρατικής νομιμοποίησης, εφαρμογής και υλοποίησης ε, προγραμμάτων αρρωγής είναι δε πάρα πολύ σημαντικό να μην σχεδιάζονται αυτά τα προγράμματα επί τη βάση υπερβολικά αισιόδοξων προβλέψεων. Ε, βάσει τροπολογία 161 του Όλε Σμιτ καλούμε το Συμβούλιο να επανεξετάσει την εμπλοκή της, ε, ε, τη συνεργασία της του και Τρόικα. Δεύτερον, για να κάνουμε άλλο ένα βήμα προς αυξημένη διαφάνεια σε σχέση με την εμπλοκή της ΕΚΤ στα κράτη-μέλη που βιώνουν χρηματοοικονομική κρίση είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να τονίζουμε όπως και το κάνουμε στην τροπολογία 112 ότι η αρχή της μη φερεγγιότητας ε, που, στην οποία βασίζεται και η αρχή της ρευστότητα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν χαρακτηρίζεται από την απαιτούμενη διαφάνεια γιατί καλύπτει και την περίπτωση όπου ε, νομικός έχει προσδιοριστεί η μη φερεγγιότητα μιας τράπεζας ή εναλλακτικά όταν όταν οι εποπτικές αρχές της τράπεζας προσδιορίζουν ότι ένα πιστοτικό ίδρυμα δεν συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπεται στο πλαίσιο για τις κεφαλαίκες απαιτήσεις. Ε, επίσης θα πρέπει ε, για να αγγιηθούμε την νομική ασφάλεια και να προωθήσουμε την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα να στηρίξουμε σχετικές τροπολογίες. Την τροπολογία 146 ζητείται από την ΕΚ να κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο τις μυστικές συμφωνίες για τα net financial assets, τα καθαρά στοιχεία των ενεργητικού ανάμεσα στις εθνικές κεντρικές τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού όπως τα κρατικά ομόλογα όπου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να έχει στον ισολογισμό τη. Όντω η ΕΚΤ πρέπει να είναι ανεξάρτητη, λέω εγώ, και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και αδιαφανή. Ε, τέταρτον, ε, για το θέμα τη επίγουσας ε, βοήθεια δρευστότητα, θα θέλαμε να παρακινήσουμε την ΕΚΤ να ενισχύσει τη διαφάνεια τη και να αποκαλύψει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανά χώρα και του όρου που ισχύουν για αυτά και τα επιτόκια και τι επιστοτικές γραμμέ. Σε σχέση με τι γραμμέ, ΕΛΑ για την επίγουσα Σα βοήθεια και το ολοκληρωμένο σύστημα των οικονομικών λογαριασμών, ε, μάλλον ε, όταν μιλάμε για την ενιαία λογιστική κατάσταση και φτάνουμε τα 603, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι τα ποσά. Ε, επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε στην ΕΚΤΕ ότι έχει αναλάβει δέσμευση νομική να κοινοποιεί όταν συνδυάζονται με τα προγράμματα τις απευθείας νομισματικές παρεμβάσεις της OMT, γιατί έτσι αυξάνεται η δημοκρατική νομιμοποίηση των προγραμμάτων του ESM. Επόμενο σήμερα σημείο. Κάποιες τροπολογίες μας ε, αποσκοπούν στο να χορηγήσουν πρόσβαση στις αγορές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και να ενισχύσουν το ρόλο τους ε, από αυτή την άποψη θα έπρεπε όσοι παίρνουν ρευστότητα από την ΕΚΤ να αυξήσουν ναι, την δανειοδοσία προς ε, τον ιδιωτικό τομέα και δεύτερον η ΕΚΤ θα πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες εφαρμογής ε, μη συμβατικών μέτρων με στόχο καλύτερες, ευνοϊκότερες ε, συνθήκες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ στην ενιαία αγορά. Κυρίως δε αν λάβουμε υπόψη ε, τα επίπεδα ανευπροηγουμένου για αρρωγή ή για και καλυμμένες επιδοτήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα. Τροπολογία 59, Σιλβί Γκουλάρ και 63 και 68, 125, 127 και 128 του Τρεμόσα μας βρίσκουν σύμφωνος. Επίσης, τροπολογία 70, Μπάλσε και 77 της κυρίας Μπατσέσκου. μακροοικονομικές προϋποθέσεις δηλαδή για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παίρνουν βοήθεια από την ΕΚΤΕ για να αυξήσουν τις δικές τους γραμμές πίστοσης προς τις ΜΜΕ σε σχέση με τις υποσχετικές της Ιρλανδίας και τα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού. Ε, περιμένουμε την αξιολόγηση της ΕΚΤΕ και τους κανόνες περί δημοσιοποίησης. Ε, ε, τέλος, Πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να ενισχυθεί το τμήμα της έκθεσης που σχετίζεται με την Τραπεζική Ένωση. Αυτό θα καλύπτει και μία αναφορά σε ένα αποτελεσματικό υπερεθνικό αποθεματικό για προμήθεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενίος μηχανισμός εξυγίανσης και ενισχυμένα πρότυπα για την κατάθεση των εγγυήσεων και τέλος αλλά εξίσου σημαντικό θα έπρεπε να αποδώσουμε σημασία σε ένα υποχρεωτικό σύστημα ε, θέσπισης ενός αξιόπιστου και καλά προσδιορισμένου πλαισίου που είναι απαραίτητο για την πραγματική οικονομία. Πρέπει επίσης να προσέξουμε τις υπερβολικές τροπολογίες. Τροπολογία 24, Λάγκερ παραδείγματο χάρη, παραπονιέστε γενικόλογα ότι είναι υπερβολικά χαμηλό το επιτόκιο. ισχύουν διαφορετικά πρότυπα ανάλογα με την αγορά και να αφισβητούμε ΕΕ το ενεύστοχο το σχόλιο ο συνάδελφος Έπινγκ ε, προσπαθεί να μας πει ότι τα προγράμματα εξαγοράς ομολόγων είναι παράνομα και χρησιμοποιεί την έκθεση. Μα ε, είναι ε, ανάρμοστο να χρησιμοποιείται η έκθεση της ΕΚΤΕ για τέτοιους ε, σκοπούς. Ε, ε, πολύ καλές συμβαστικές προτάσεις και με τις ανταλλαγές απόψεων ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συνενετικές λύσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε να μου πείτε άμα θέλετε το λόγο και πριν ξανακούσουμε τον εισηγητή. Πολ, μπορείς να αρχίσεις να κυνηγά αυτούς που θα χρειαστούμε για τα σημεία 15 και 16 της ημερησίας διάταξης. Γιατί δεν θέλω άλλη διακοπή. Ντανίτα Χούπνερ, Νταμίτσι, εγώ είμαι εδώ, Φιλίπ Λάμπερς και Γιώργιν Κλούτε. Γιατί ακολουθούν μετά την έκθεση και η Σουίμπορν. Βρείτε και τους σκιώδη σας λοιπόν για το σημείο 16 και να έρθουν νωρίτερα από ό,τι είχαν προβλέψει. Να είναι στην αρχή να έρθουν νωρίτερα πριν αρχίσει η συζήτηση του θέματος. Μπορείς να μιλάς για μισή ώρα, Τζάνι. Μα όχι δέκα δευτερόλεπτα. Θα τα πω γρήγορα. Ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους. Τις ήξερα τις θέσεις, γιατί ξέρω και τις πρωτοτροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό ειδικά αυτά τα σημεία της διαφάνειας ε, και άλλα. Αλλά την ε, Πέμπτη το πρωί θα τα ξαναδούμε και θα δούμε με ποιο τρόπο θα καταλήξουμε στην πλέον ενδεδειγμένη έκθεση που να αντανακλά τις πλειοψηφικές θέσεις της Επιτροπής μας. Okay, thank you very much. Um, the time... Ευχαριστώ πολύ χρονοδιάγραμμα. Θα ψηφίσουμε 4 και 5 Νοεμβρίου προσπαθώντας να το πάμε το θέμα στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, όχι όμως μέχρι τις 4 και 35 που έλεγε το πρόγραμμα. Θα πρότεινα ανταυτού να κάνουμε ένα μικρό διάλειμματάκι μέχρι ε, στις 4 και 4, δηλαδή 20 λεπτά πιο νωρί και ίσως έτσι καταφέρουμε να τελειώσουμε και πιο νωρί τη συνεδρίαση συνολικά. Λεζον έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό. Απάντηση, όχι, όχι. Αλλά δείτε πόσοι συνάδελφοι είναι παρόντες. Φοβάμαι ότι αν τους δώσουμε 20 λεπτά ίσως να εξαφανιστούν και οι αναπομείναντες συνάδελφοι. Θα ήταν λίγο λυπηρό τελικά να το συζητήσουμε οι δυο μας το θέμα. Όχι ότι... Δεν δηλαδή, δε, δε ξέρω, ίσως να μην είναι και τόσο λογικό να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα. Πρόεδρος, ένα τέταρτο είπα να κάνουμε διάλειμμα, όχι τρία τέταρτα και ε, ρώτησε αν είναι δυνατόν να βρεθούν οι ε, συνάδελφοι που θα έπρεπε να είναι παρόντες για τα σημεία 15 και 16 της ημέρας διάταξης. Τώρα, αν διαφωνείτε να μην κάνω διάλειμμα, αλλά κάποιοι από εμά είμαστε παρόντε. Άλλοι δεν είναι όμως. ένα πρόβλημα συμφωνική και να το συζητήσουμε τώρα, αλλά ίσω υπάρχουν συνάδελφοι που να θέλουν να εκφράσουν την άποψή του πάνω σε αυτό το ζήτημα ανακάμψη και τη εξηγένσης για τα μειοπιστωτικά ιδρύματα. Στην ημερήσια διάταση έλεγε 4 και 35 και προτείνω να το κάνουμε 4 και Τέταρτο έτσι ώστε οι συνάδελφοι να έρθουν στην αίθουσα. Και επίση να αναζητήσουμε και εκείνου που θα πρέπει να μιλήσουν για του λογαριασμού πληρωμών. Γιατί διαφορετικά απλώ θα καθόμαστε και θα κοιτάμε τον καιρό έξω. Ευελπιστώ ότι οι βοηθοί έχουν ήδη αρχίσει να στέλνουν SMS στα μέλη του Κοινοβουλίου. διαλυματάκι 5-10 λεπτών, εκτό αν έχεις οποιαδήποτε άλλη ιδέα. Ευχαριστώ να την ακούσω. Okay, right, let's, let's resume. We've gathered together. Ωραία, ξαναρχίζουμε. Έχουμε τους βασικούς παίκτες για την έκθεση της ΚΕΙ. Ο Λεωνάρδο δεν μπορεί να έρθει για τους σοσιαλιστές. Ε, θα μας έχει στείλει, ε, μας έστειλε τις σημειώσεις του γραπτός, αλλά δεν υπάρχει κανένας βουλευτής των σοσιαλιστών για να τις διαβάσει. Μπορεί να τις διαβάσω εγώ. Αφήστε που είναι και στα Ιταλικά. Έλο πάντων θα, το, θα διασχίσουμε αυτή τη γέφυρα όταν φτάσουμε εκεί ή θα ξεπεράσουμε το σκόπιλο όταν πέσουμε πάνω. Okay. Ευχαριστώ. Εν γέννη υπάρχει μεγάλη επικάλυψη ανάμεσα στις τροπολογίες που υπέβαλαν οι πολιτικές ομάδες και παρότι δεν υπάρχει επικάλυψη ανάμεσα σε μεμονωμένες τροπολογίες ε, εγώ ως συγγήτρια μπορώ να υποστηρίξω τη συντριπτική πλειοψηφία των ε, τροπολογιών διότι συνιστούν πραγματική ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με την αρχική έκθεση. Δεδομένου του επίπεδου συνένεσης λοιπόν για όλες αυτές ε, τις τροπολογίες την περασμένη εβδομάδα και έστειλα ένα πρώτο σετ τροπολογιών που βασίζονται σε αυτές. Ε, οι σκιώδεις έχουν λάβει αυτό το σετ τροπολογιών, αλλά είναι στη διάθεση όλων. Όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχουν διάφοροι τομείς όπου δεν είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου ε, ποια κατεύθυνση θέλουν να ακολουθήσουν οι συνάδελφοι και μεταξύ άλλων σχετίζονται αυτά με τις τροπολογίες του κ. Ντομινίτση και καλό θα ήταν κάποιος να μας διαφέρει φώτιζε για κάποιες τροπολογίες γιατί ε, έχω μπερδευτεί για κάποιες και δεν ξέρω ακριβώς ποια κατεύθυνση προτείνουν να ακολουθήσουμε. Οι δικές μου τροπολογίες για την εκθεσή μου ήταν περιορισμένο αριθμό. Προσέθεσα πληροφορίες σε σχέση με δημοσιοποιημένες ε, πληροφορίες, ε, πληροφορίες μάλλον που δημοσιεύτηκαν μετά την έκδοση του πρώτου σχεδίου και υπάρχει μία προφανής αμφισημία ε, μέσα στην έκθεση και αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε. Μου το υπέδειξαν συνάδελφοι. Υπάρχουν και θέματα διατύπωσης που ρυθμίζουμε μέσα από τις τροπολογίες. Ας καλύψω κάποιους κάποια ζητήματα τακτοποίησης και χτενίσματος ε, στον ασφαλιστικό τομέα παραδείγματος χάρη. Όπως είπαμε και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι περιορισμένα αυτά που λέμε για τον ασφαλιστικό τομέα αλλά έχουμε από την ε, Διεθνή Ένωση Εποπτών του Ασφαλιστικού Τομέα έχουν, έχουν, έχει εκδώσει δύο εκθέσεις και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να γίνουν και άλλες έρευνες στον τομέα προτού εμείς νομοθετήσουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρόωρο ακόμη ε, από πλευράς ε, ε, συστημικής σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο Έχουμε εντοπίσει κάποιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι όλες ε, συστημικά σημαντικέ και άρα επικίνδυνε. πρέπει να, ε, να φροντίσουμε να προχωρήσει και η δουλειά για το Omnibus 2 και για τη Φερεγγιότητα 2 πρωτού εμείς προχωρήσουμε. Θέλω να προδικάσω την έκβαση δηλαδή με την έκθεσή μου. Ε, τώρα, για τις δικές μου τροπολογίες ε, συνεχίζω, προσπάθησα να ε, για τα σχέδια εξυγίανσης ε, να πω ότι τα όσα κεντρικά αποθετήρια λειτουργούν με τραπεζική άδεια πρέπει να καλυφθούν από την BRRD κάποια μέλη της Επιτροπής ε, θέλησαν ε, να αναφέρουν συγκεκριμένα ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες σε περίπτωση κρίσης. Πέρα από το διακανονισμό είναι όντως καταλητική σημασία, αλλά ε, έχουμε και το, τις core services, τις βασικές υπηρεσίες των κεντρικών ε, αποθετηρίων τίτλων και ο ΟΣΚΟ παραδείγματος χάρη ε, έχει κέρυες τέτοιες υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε στον προσδιορισμό των βασικών υπηρεσιών των ΚΑΤ. Ε, υπάρχουν και κάποιες άλλες απόψεις όπου είναι μάλλον πιο αποκλίνουσες ε, οι απόψεις ε, όταν μιλάμε για τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους και την εξυγίανσή τους. η CPSS, η ΟΣΚΟ δημοσίευσε την σχετική έκθεση και νομίζω ότι ε, όλοι τη διάβασαν γιατί αναγνωρίζω τη διατύπωση στις τροπολογίες που κατέθεσαν οι σκιώδεις. Επιθυμούμε διεθνή σύγκληση και ε, διασυνοριακής φύσης για τους ε, κεντρικούς αντισυμβαλωμένους, ε, για τα κάτι και άλλες υποδομές. Δηλαδή πρέπει να έχουμε διαρκώς κατά νου αυτή την πτυχή και έχουμε καταθέσει σχετικέ τροπολογίες. Επίσης, κατέθεσα τροπολογίες για την ανάκαμψη και εξυγίανση των CCP των αντισυμβαλωμένων, γιατί εκεί μου φαίνεται ότι έγκυται οι περισσότερες αμφισημίες και όλα τα προϊόντα που εκαθαρίζει ο κεντρικό ενός πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο εξυγίανσης, λέω. Όμως αναγνωρίζω ότι μπορούμε να δώσουμε ιδιαίτερη ε, σημασία στα προϊόντα που έχουν εντολή για κεντρική εκαθάριση, γιατί παραδοσιακά δεν περνάνε από τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και μιλάμε για διαφορετικούς παίκτες ε, της αγοράς και ενδεχομένως να χρειαστεί να συνεκτιμηθούν και διαφορετικοί παράγοντες. Ε, θα δούμε αν όλα τα προϊόντα, δηλαδή όλα τα προϊόντα θα αναγράφονται ε, μέσα στο σχέδιο εξυγείας, ανάκαμψης και εξυγείας, αλλά για κάποια υπάρχει συγκεκριμένη εντολή για κεντρικό διακανονισμό. Ε, τώρα για το Ταμείο Αθέτηση Υποχρεώσεων, Default Fund, ε, εάν ε, λάβουμε υπόψη τη CRD και το ΕΜΙΡΕ και την ε, έλλειψη εγγυήσεων που τόνισαν πολλοί, ε, τι μας λένε οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι, ότι προσπαθούν να αποφασίσουν πώς ακριβώς θα καλύψουν το θέμα της έλλειψης εγγυήσεων, γιατί αυτό τους δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εάν τώρα υπάρχει στα στο πλαίσιο ενός κεντρικού αντισυμβαλόμενου δυνατότητα πολλαπλών περιθωρίων τότε ε, ενδεχομένως να ανακύψουν συγκρούσεις ε, συμφερόντων. Μπορεί να έχετε ένα μικρό ταμείο αθέτηση υποχρεώσεων ε, που δεν θα καλύπτει τις ανάγκες σε περίπτωση κρίσης. Οπότε πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Συνιστά αυτό σύγκρουση συμφερόντων ή μήπως στο επόμενο αναθεωρημένο σχέδιο του σχεδίου ανάκαμψης και εξυγίανση ε, θα έπρεπε ε, να καλύφθουν. Υπάρχει αυτό το trigger point ανάμεσα στην ανάκαμψη και στην εξυγίανση ε, για τη μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο. Δηλαδή αυτό το trigger point, το σημείο ενεργοποίησης δηλαδή, απασχόλησε τους σκιώδες στην τελευταία συνεδρίαση που κάναμε. Αυτό που θέλουμε εμεί είναι η αρχή εξυγίανση να έχει την εναλλακτική να κινηθεί πέρα από ε, τον κανονισμό ΕΜΙΡ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν εκεί οι αντισυμβαλόμενοι στο δικό τους σχεδιασμό, δηλαδή στη δική τους διαχείριση, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να βασίζονται στο ότι μπορούν να έχουν επιπρόσθετα εργαλεία ανάκαμψης, ε, παραδείγματο χάρη ε, να ενισχύσουν το Ταμείο Εξυγίανσης, αλλά πέραν αυτού να μπορεί και η αρχή να παρέμβει το νωρίτερο δυνατόν, εάν κρίνουν ότι είναι σημαντικό είτε για να προστατεύσουν ε, τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, να προστατεύσουν γενικότερα την αγορά. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να πούμε ότι ο αντισυμβαλόμενος με, ε, το αντισυμβαλόμενο μέρος, κανένα αντισυμβαλόμενο μέρος στην κρίση του 2008 δεν ακούμπησε ε, το Ταμείο Αθέτηση Υποχρεώσεων. Οπότε καταλαβαίνουμε και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν μιλάμε για φυσιολογικά σενάρια, μιλάμε για ακραίε καταστάσεις που ακόμα ακόμη δεν έχουμε βιώσει και γι' αυτό θα ήθελα οι αρχές εξηγένσης να έχουν πολύ μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών να έχουν τις ε, αρμοδιότητες τους ε, πέρα από τις διατάξεις περιαθέτησης υποχρέωσεων του ΕΜΙΡ και ξαναλέω η λειτουργική συνέχεια είναι το πλέον σημαντικό για μένα, δηλαδή να εξασφαλίζεται μία συνέχεια και να έχουν περιθώριο ελιγμών. Ε, για να χρησιμοποιήσουν τις αρμοδιότητες. Η αρχή εξυγίανσης ε, επίσης, ε, ξαναλέω, υπάρχει αυτό το trigger point, σημείο ενεργοποίησης. Εάν απειλούνται περιουσιακά στοιχεία πελατών, τότε πρέπει να εμπλακεί η αρχή για να εξασφαλίσει η ισότιμη μεταχείριση όλων των πελατών και όλων των ταμείων που έχει, συγγνώμη, κεφαλαίων που έχει ο αντισυμβαλόμενος. Γιατί υπάρχουν τα εκαθαριστικά σκέλη, αλλά δεν συνδέονται ε, άμεσα οι αντισυμβαλόμενοι με τους πελάτες των εκαθαριστικών μερών. Οπότε ε, όταν ε, έχουν προσφογραφεί διατάξεις διακυβέρνηση, ε, οι πελάτε δεν καλύπτονται και αυτό είναι το πιο ρηψοκίνδυνο σε περίπτωση κρίση, όταν δηλαδή τα στοιχεία ενεργητικού θα πέσουν στα χέρια κάποιων που καμία σχέση δεν έχουν με τι διατάξει που δεσμεύουν τα αντισυμβαλώμενα μέρη. Γι' αυτό σα μιλάω για τα περιθώρια. Και ότι το, αυτό το σημείο ενεργοποίησης χρειάζεται για τα περιουσιακά στοιχεία των, των πελατών. Όμως αυτό προποθέτει ότι υπάρχει επιμερισμός ε, στην ιεραρχία των ζημιών από πλευράς του κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ε, ε, είναι μια γραμμή άμυνας για τα εκαθαριστικά μέλη. Τα εκαθαριστικά μέλη, αν δεν μπορούν να υποστηρίξουν πλέον το διακανονισμό και άρα πρέπει να μετάσχουν οι πελάτες τους, τότε η αρχή εξηγένσης πρέπει να κάνει το αρμπιτράζ. Ε, τις επόμενες εβδομάδες ε, θα εξελιχθούν οι συζητήσεις, αλλά πάντως ε, από ό,τι είδα στις τροπολογίες ακολουθούμε πάνω κάτω τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ότι χρειαζόμαστε μια ευρεία συνενέση τόσο ώστε να είναι ηχηρό το μήνυμα που θα περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μας ενδιαφέρει η προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και να μεριμνήσουμε ώστε να γίνει κατανοητό πως τα κεντρικά συμβαλόμενα μέρη δεν, είναι, δεν έχουν στη δική τους ιδιοκτησία τα ε, περιουσιακά στοιχεία των πελατών. Ευχαριστώ πολύ και ερχόμαστε στους κοιόδης ηγητές από το ΕΛΚ, η κυρία Ντανούτα Χούβνερ. Ευχαριστώ πολύ Σάρον. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη αλλά θα πρέπει να φύγω γιατί είμαι και σε άλλη ε, επιτροπή ε, που πρέπει να πάω. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Κέι, γιατί έκανε ε, πολύ καλά τους συμβαστικές προτάσεις μετά τη συνεδρίαση των σκιωδών. Πραγματικά ελπίζω να βρούμε συμβασμούς και για άλλα στοιχεία της έκθεσης. Θα σας πω εγώ πώς ε, ερμηνεύω τους συμβιβασμούς και διορθώστε με ασφάλω. Οι συμβιβασμοί τονίζουν ε, ότι η ανάκαψη και τα ε, σχέδια ε, διάσωση ή εξυγίαση θα πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με το πρόκειται για τράπεζα, για ασφάλεια, ε, για CCP, για τους συμβαλωμένους και ανάλογα με τη φύση του Ιδρύματος. Υπάρχουν κάποια σημεία ε, στη χρηματαγορά και κάποια στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές. Ακριβώς ε, αν πτωχεύσουν λοιπόν ή αν κλείσουν αυτές οι εταιρείες ε, θα είναι πάρα πολύ ε, σοβαροί οι κραδασμοί. Και το σχέδιο εξυγίανσης νομίζω θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των διαφόρων αρχών. Εάν ένας όμιλος έχει υποκαταστήματα σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, τι γίνεται με τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για εκείνους που έχουν άδεια λειτουργία ως τράπεζα ε, για να ενταχθούν στο σύστημα ανάκαμψης και ε, εξυγίασης τραπεζών. Και σε ό,τι αφορά το CSD, έχω την αίσθηση ότι ενώ αρχικά η έκθεση ε, θέλει να διαφυλάξει τη βασική λειτουργία διακανονισμού, τώρα μιλάει και για άλλες βασικές υπηρεσίες του CSD και αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει διάφορες λειτουργίες και υπηρεσίες. Επίσης, υπάρχει γενικότερη αντιμετώπιση και συμπερίληψη του τομέα των ασφαλιών οι ασφαλιστικές εταιρείες ε, ε, έχουν ε, διάφορα στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη φεραγγιότητα 2, αλλά και πέρα από το διακανονισμό του 98 για τη σωστή εξυγίαση και ανάκαμψη για συστήματα πληρωμών. Συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα που μπορεί να μην καλύπτονται γιατί ακόμα δεν έχουμε βρει συμβιβασμούς. Ελπίζω να προχωρήσουμε κατά τη ε, συνεδρίασή μας την άλλη εβδομάδα για να προχωρήσουμε να τα λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Και ιδιαίτερα και την αξία που προέρχεται από τους πελάτες και στο clearing, ε, στις καθαρίσεις και ε, ιδιαίτερα στις διάφορες ε, τάξεις ε, στοιχείων ενεργητικού, τα διάφορα είδη στο CCP και το σημείο ακριβώ που δρομολογείται η εξέλιξη, το trigger point που πυροδοτείται και ένα τελευταίο που για μένα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να βρω το συμβιβασμό έχει να κάνει με το αν συμμετέχουν εθελοντικά ε, οι οργανισμοί εκαθάρισης ε, και οικονομικά. Και ποιος θα πληρώνει δηλαδή, θα πληρώνουν οι πελάτες ή οι ίδιοι. Πάντως ε, καλό είναι που προχωρούμε προς μια κατεύθυνση που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και κατανοούμε και τις δυσκολίες και τις προκλήσεις σε αυτό το κλάδο. Ευχαριστώ πολύ την για όλη τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Thank you, Ευχαριστώ, Ντανούτα. Όντω είναι δύσκολο όταν πρέπει να προεδρεύει και σε άλλη επιτροπή να έρχεσαι εδώ να τα λες. Ε, δεν βλέπω ε, αν θέλει κανένα να διαβάσει τα, τις σημειώσεις του Λεωνάρντο. Εγώ είμαι σκιώτης από την ομάδα μου, να πω και εγώ τα δικά μου. Ε, ευχαριστώ την Κέι για την έκθεση. Δεν έχω κάνει πάρα πολλέ τροπολογίε και ήταν λογικό γιατί εσύ πολύ σωστά τα λες στην αρχική σου ε, παρουσίαση, οπότε δεν χρειάστηκε να κάνω τροπολογίες. Ε, αν θέλουμε να κάνουμε μια ενιαία νομοθεσία, αυτό αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καλύπτει όλα τα μη πιστοτικά ιδρύματα, όλα τα μη τραπεζικά δηλαδή. Αυτό θα χρειαζόταν πολλά νομοθετήματα γιατί δεν χωράει σε μία νομοθεσία όλος αυτός ο τομέας και ο κλάδος. Θα πρέπει να παραμείνουν κάποιες κρίσιμες λειτουργίες ε, σε καιρούς μεγάλης πίεσης και όλες οι τροπολογίες με τον ΑΒ τρόπο προς τα εκεί στοχεύουν. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να λάβουμε υπόψη τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και προαπαιτήσεις το, ε, ε και τον Όσκο και ε, κάποια άλλα διεθνή ισχύοντα. Ε, εμείς μπορεί να θέλουμε όμως λίγο πιο λεπτομερή και πιο λεπτή ρύθμιση, γιατί αυτά είναι κάπως αδρές ε, γενικές κατευθυντήριες γραμμές και ρυθμίσεις. Εμείς θέλουμε ίσως πιο πολλές αποχρώσεις. Δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με τα διεθνώς ισχύοντα. Ίσως θέλουμε κάποια διευκρίνηση. Ε, στην τροπολογία μου 80 αναφέρω μερικά στοιχεία ε, για την κρίσιμη λειτουργία και πώς ε, διευρύνεται το πλαίσιο των λειτουργιών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τι συμβαίνει και όχι πάντα οι λεπτομέρειες για το πώς θα φτάσουμε εκεί. Η CCP αντισυμβαλόμενη είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι πολύ σημαντικό τη μείωση κινδύνου πτώχευσης από την κεντρική εκαθάριση και από κάποιον αντισυμβαλόμενο. Δεν προστατεύονται πάντα από το κλείνει την εκαθάριση όταν οι ε, αντισυμβαλόμενοι ε, πτωχεύουν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι αρχές των συμβατικών υποχρεώσεων και όχι πώς τα κράτη-μέλη μετακυλίουν ε, στους πελάτες τους τις ή τα μέλη μετακυλούν μάλλον στους πελάτες τους τις απώλειες. Για κάτι που δεν φταίνε και ε, που είναι ε, σφάλμα η πετιότητα των CCP, ε, των αντισυμβαλωμένων. Πού είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ανάκαμψη και την εξυγίαση εξυγένση γίνεται εφόσον εξαντληθούν όλες άλλες οι πριν την πτώχευση και ε, όλα τα άλλα που ε, αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατευτεί το σύστημα, έτσι, το ring fencing. Αλλά σε ό,τι αφορά την εξυγένση των τραπεζών, ε, την ανάκαμψη, Υπάρχουν και επεμβάσεις που μπορεί να μην ακολουθούν 100% το σχέδιο ανάκαμψης, γιατί δεν μπορεί πάντα ένα προς ένα να αντιστοιχεί η πραγματικότητα στο σχεδιασμό. Χρειάζεται κάποια στοιχειώδης ευελιξία, στο βαθμό που εξηγείται αυτή, όμως και μπορεί να υποστηριχθεί. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει ένα σχέδιο ανάκαμψης και εξυγίανσης, αλλά από εκεί και πέρα τι και στον τριμερή διάλογο για την εξηγέση των τραπεζών. Καμιά φορά ακούμε διάφορες φωνές για να μην πω θορύβους από πλευρά Συμβουλίου που μάλλον υποτιμούν τη σημασία των σχεδίων ανάκαψης. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένας χάρτης, ένα φύλλο πορείας, ένας μπούσουλας για τους επενδυτές να ξέρουν τι τους περιμένει. Και αυτό σημαντικό δεν είναι. Και όταν φτάσουμε στην εξυγίαση, στη διάλυση, ε, απλούστατα θα πρέπει να γίνεται ανάληψη όλων των θέσεων. Να δούμε και το θέμα λοιπόν της διαλειτουργικότητας και πώς μπορεί να γίνει αυτή η ανάληψη εξ αγορά. Αν υπάρχουν διατάξεις για την πρόσβαση. Δεν μπορεί απλούστατα να περάσει κάποιος έναν άλλο αντισυμβαλόμενο. Ε, από ένα πτωχευμένο. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ε, ξαπατούμε κάπως ή ε, απογοητεύουμε το κοινό. Είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα και να ξέρουμε τι γίνεται σε περίπτωση πτώχευσης. Τώρα για τις ασφάλειες, όντως κάτι πρέπει να κάνουμε και για αυτές τις εταιρείε για την ανάκαμψή τους και την εξυγένσή τους. Δεν πιστεύω ότι αυτό όμως μπορεί να μπει κάπου σε ένα μεγάλο πλαίσιο εξηγένσης που να καλύπτει τα πάντα στις ασφαλιστικές εταιρείες αυτή η προσπάθεια είναι πιο δύσκολη από τις δράπεζες. γιατί το, το παθητικό τους ε, και τα στοιχεία ε, και τα χρέη τους και όλα αυτά είναι κάτι πολύ μακροπρόθεσμα, έχουν μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες και δεν μπορούμε έτσι ελαφρά την καρδία να το διεκπεραιώνουμε. Κάποιος τρόπος πρέπει να βρεθεί. Στη φερεγκιότητα Δύο προσπαθήσαμε ε, να το κάνουμε, αλλά μάλλον να βάγει σε αυτή η προσπάθεια και στην περίπτωση της εξυγίανσης και ανάκαμψης των τραπεζών έχουμε και το πρόβλημα της διασυνοριακής ε, μεταφοράς στοιχείων ενεργητικού και για τα CSD όπως προτείνατε μπορεί κάποια στιγμή να πείτε ότι εντάξει όταν υπάρχει ένα πρόβλημα μπορούμε να βρούμε κάποια λύση, να χρησιμοποιηθούν ορισμένα άρθρα ή κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού, asset managers, ε, έχουν διαχωριστεί αυτοί και μπορεί να μην είναι πάντα οι ίδιοι ε, που διαχειρίζονται τα στοιχεία. Δηλαδή όταν καταρρεύσει κάποιος ε, διαχειριστής να μην παίρνει μαζί του και τα στοιχεία ενεργητικού. Να υπάρχουν κάποιοι θεματοφύλακες ε, και να παρακολουθούμε τι γίνεται ε, σε κάποιον διαχειριστή. Γιατί όταν ένας μεγάλος τέτοιο παίκτη καταρρεύσει, δεν θα πρέπει να παίρνει μαζί του και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και να χάνονται. Κάποια στιγμή να υπάρχει μια εξαγορά και τελικά ενδεχομένως να μην χάνονται αυτά τα στοιχεία. Αυτές ήταν οι δικές μου θέσεις και οι τροπολογίες που θα κάνω και ελπίζω να τα ξαναπούμε στους και οδησηγητές, αλλιώς θα στείλουμε ε, τις σημειώσεις. Αν χρειαστεί να είμαι σε κανένα τρίγλογο ή τίποτα τέτοιο. Ε, ε, τους πρασίνους τώρα, Φιλίπ Λάμπερς. Thank you, ε, Ευχαριστώ, Σάρων. Μακάρι να βρεθούμε στη συναντήσει συναντήσεις οδόν και εσύ και εγώ και η Αλλά από ό,τι φαίνεται τελικά δεν θα ε, συνεργαζόμαστε με τη Βίκη σε κάθε έναν από του φάκελους. Να ορίστε που θα συνεργαστούμε και με εσένα και με την Κέι. Για να δούμε πώς θα πάει. Δεν εννοώ ότι υπήρξε κανένα πρόβλημα στη συνεργασία με τη Βίκη. Λοιπόν, κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα με ανησυχεί το γεγονό ότι δημιουργούμε ένα νομοθετικό πλαίσιο για τις τράπεζες το οποίο δίνει ε, πλεονέκτημα σε ορισμένα μη πιστοτικά ιδρύματα τα οποία ανταγωνίζονται τις τράπεζες και θα πρέπει νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ε, δράση, όχι να αναμένει τις ε, κινήσεις ε, των κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, η οδηγία BRD δεν θα έπρεπε να παρακαμφθεί από τα μη πιστοτικά ιδρύματα, BBRD, γιατί αυτό θα υπονομεύσει τη γενικότερη αποτελεσματικότητα του συστήματος εξυγένσης παρόλο που σε γενικέ γραμμές εγώ δεν υποστηρίζω αυτή την ε, λογική του ισότιμου ανταγωνισμού, εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το προσέξουμε. Τώρα, δεν είναι σκόπιμο να ε, βάλουμε στο, όλα μαζί ε, ιδρύματα που είναι τράπεζες, ιδρύματα που δεν είναι πιστοτικά στο ίδιο πακέτο. όσον αφορά τη εξηγήση των CSD και των CCP και των αντισυμβαλωμένων αυτά τα αυτοί οι αντισυμβαλόμενοι είναι ένα μέρος του συστήματος, επομένως οδηγούν σε συστημικό ρίσκο. Το γεγονό ότι ακόμα δεν είχαμε κάποια κρίση με κάποιο τέτοιο ίδρυμα δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί και στο μέλλον. Δεν υπάρχει ε, χρηματοδοτικό μέσο ε, για τα CDS το οποίο ε, θα φέρνει υπέρογκα ποσά στην EAG χωρίς ποτέ να κοστίσει τίποτα. Τελικά οι φορολογούμενοι θα κληθούν να το πληρώσουν αν συμβεί κάτι τέτοιο. Επομένως, σε συγχαίρω για την προετοιμασία. Πέρα από το trigger, το σημείο εκκίνησης νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τώρα, σε αυτό που είπατε για το trigger. Ήταν μια συζήτηση που την είχαμε και σε σχέση με την BRRT για την εξήγηση των εντρωμάτων. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στη διακριτική ευχέρεια αφενός και την δυνατότητα πρόβλεψης, την προβλεψιμότητα δεν πρέπει να φτάσουμε στο ένα άκρο, δηλαδή να περιμένουμε ότι αυτό, ο, ο, ο, ο τρόπος ε, αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων θα ήταν μια συνταγή, ένα αλγόριθμο που θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα υπολογιστή. Αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να φτάσουμε και στο άλλο άκρο, ε, ε, μια αριθμιστική αρχή να έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια και να της δώσουμε τη δυνατότητα να λάβει αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε προβλήματα συνολικά σε μια ολόκληρη κοινωνία και οικονομικά προβλήματα. Επομένως πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Δηλαδή ε, το, το, το αίτημα για προβλεψιμότητα αφενός και την ύπαρξη διακριτικής ευχέρειας αφετέρου στην ξύγερση και καθάριξη. Νομίζω για να το πετύχουμε αυτό σημαντικό θα ήταν οποιαδήποτε παρέκκληση από το σύνηθες να ε, δικαιολογείται και να, να, να αιτιολογείται όταν αυτή η παρέκκληση μειώνει το συνολικό κόστος της εξυγίανσης, το κόστος που υπομίζεται η ε, κοινωνία, ο φορολογούμενος. Με αυτόν τον τρόπο τελικά το κράτος, η ρυθμιστική αρχή ε, προστατεύει τα συμφέροντα της κοινωνίας συνολικά. Εάν αυτό σημαίνει ότι θα αναλάβουν μεγαλύτερο κόστος οι ε, επενδυτές εκείνου του συγκεκριμένου ιδρύματος, ας έχει αφού θα προστατευτεί η κοινωνία συνολικότερα. Χρειάζεται να ενισχύσουμε το σύστημα που δημιουργήθηκε με το πακέτο φερογιδότητα 2. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αντίσταση από ε, μέλη του, του κλάδου, ε, για παράδειγμα στον τομέα της, ε, του ευμετάβλητου της αγοράς μας ανημέρωσε αυτές και ο κ. Βάγκη. η εξυγίανση μιας ασφάλειας ζωής είναι κάτι διαφορετικό από την εξυγίανση ενός ιδρύματος από το EAG, ας πούμε, που ασχολείται κυρίως με την ασφάλιση παραγόγων ή χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στη μία περίπτωση μπορούμε να προβλέψουμε το γεγονό ότι πηγαίνουμε πάνω σε ένα παγόβουνο και πάμε να το χτυπήσουμε Ενώ στην άλλη περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη, υπάρχει διάχυση των εξουσιών και δεν είναι τόσο απλό να, γίνει, ε, να, να ληφθούν οι αποφάσει για την εξυγίανση. Στα τροπολογίες 7, 8, 21 και 28 διαπιστώσαμε ότι ακολουθήσατε τις προτάσεις μας και σας ευχαριστώ για αυτό δεν φαίνεται να ακολουθήσατε την πρόταση. που αφορούσε τους αντασφαλιστές. Από ό,τι φαίνεται δεν θα επιθυμείτε η Επιτροπή να εξετάσει το θέμα αυτό των αντασφαλιστών. Για τις σκιώδεις τράπεζες τώρα. Όπως γνωρίζετε, ένα σημαντικός ε, όγκο των τραπεζικών συναλλαγών κατευθύνεται προς τις χειώδεις ε, τράπεζες και αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις, θα δημιουργήσουμε προβλήματα στη λειτουργία του κλάδου εάν τελικά επιβάλλουμε ε, απαιτήσει στι επίσημε τράπεζε οι οποίε δεν θα αφορούν τι σκιώδει τράπεζε γιατί στην πραγματικότητα αυτά τα ιδρύματα έχουν, εκτίθενται στο ίδιο βαθμό κινδύνου. Άρα πρώτον θα έπρεπε να ε, καθορίσουμε με σαφήνεια ποια είναι αυτά τα μη πιστοτικά ιδρύματα και δεύτερον να καθορίσουμε ένα σαφές ε, καθεστώς και διαδικασία εξυγίανσης. Για την 109 και την 110 θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του εισηγητή. Και Ένα στοιχείο που ίσως συχνά ξεχνάμε, μάλλον λόγω φόρτου εργασίας, είναι το εξή. Προσπαθούμε να μάλλον εξετάζουμε κάθε στοιχείο του χρηματοπιστωτικού τομέα ξεχωριστά. Αλλά το συστημικό ρίσκο πολύ συχνά προκύπτει από την αλληλεπίδραση αυτών των μερών του συστήματος. Άρα θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εποπτείας της χρησιμοπιστωτικής οράς και αυτό προσπαθούμε να το εκφράσουμε στην ε, ε, τροπολογία 138 να δημιουργήσει ένα σύστημα ε, εποπτείας του συστημικού ρίσκου που προκύπτει από το δίκτυο των αλληλεπιδράσεων, δηλαδή να μελετήσει ακριβώς πώς οι συλλαλλαγές μεταξύ αυτών των στοιχείων του συστήματος δημιουργούν κίνδυνο. Φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, δηλαδή να αποφύγουμε να χρειαστεί να φτάσουμε στην εξυγίανση και την ανάκαμψη, αλλά χρειάζεται να έχουμε τα μέσα στην διάθεσή μας για να φτάσουμε εκεί. Ε, λοιπόν να συμμετάσχουμε στη συζήτηση εν ώψη του τριμερούς διαλόγου. Γιώργη, θέλεις το λόγο? Όχι. Έχουμε στείλει γραπτός ε, σχόλια, ε, αλλά ασχολούμαι με τη δική μου την έκθεση. Τώρα ναι, ναι, θα φτάσουμε και σε αυτό λέει η κυρία Μπόλς. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Εγώ θα καταχραστώ τη θέση μου ε, προ, της Προέδρου και θα προκαλέσω πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτά που ε, καλά κάνουμε και λέμε ε, αυτά που λέει ο Λάμπερτς ότι η ίδια έκθεση, ίδιος κίνδυνος αλλά όταν είναι συστημική σημασία ε, το ίδρυμα είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Σε μία τράπεζα, κατά τη διαστολή με μία σκιώδη τράπεζα και όλα αυτά είναι συνάρτηση τη φύση των δραστηριοτήτων της ε, σκιόδους τράπεζας ε, γιατί είναι... Εξαρτάται πώς επηρεάζεται δηλαδή η κοινωνία ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων και θα πρέπει και αυτό να το συνυπολογίσουμε ούτως ώστε να είναι αναλογικά τα μέτρα με τη φύση ε, των Ιδρυμάτων και τη συστημική τους ε, σημασία. Αυτό ήθελα να πω. Okay. Θέλεις να κάνεις ε, τις τελικές παρατηρήσεις. Ναι. Για αυτό που είπε ο Φιλίπ, οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το κείμενο, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό και έτσι κι αλλιώς θα ψηφιστεί ξεχωριστά το θέμα της αντασφάλισης είναι ολόκληρος τομέας, ξεχωριστός κλάδος ε, που δεν έχει και καμία ε, σχέση. Δεν λέω ότι δεν είναι κρίσιμος, απλώς αν θέλουμε να μπει σε αυτή την έκθεση, όχι. Αυτό το δούμε στις τροπολογίες. Και κάποιες άλλες τροπολογίες χρειάζονται ε, κάποιες προσθήκες και τα λοιπά. Προσπαθούμε λοιπόν να επικεντρωθούμε σε κάποια θέματα που ανήκουν σε αυτή τη θεματική ενότητα και όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός. Ε, ως προς τις ομοιότητες εδώ και τη συνέχεια ε, του κλάδου και των υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει όλους σύμφωνους πέρα από πολιτικές ομάδες και είναι κρίσιμο να πούμε ότι είναι διαφορετικά τα εργαλεία ανάλογα με το πρόβλημα. Αν το πρόβλημα ήταν στη διαχείριση και στη δίκηση είναι τελείως διαφορετικό ε, από το... Ε, δεν θα, μπορεί να πτωχεύσει ένας φορέας, ένας ε, ε, διαχειριστής σε μια αγορά χωρίς να καταρρεύσει όλος ο κλάδος. Και για την ορολογία, ε, Πρόεδρε, για οποιαδήποτε διαφάνεια ε, που χρειάζεται η ε, κάθε ευελιξία. Υπάρχουν πολλοί αντισυμβαλόμενοι που λένε ότι δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα. Συμφωνώ, αλλά μπορείς να προβλέψεις πάρα πολλά. Και μπορεί να υπάρχει ένας ε, χάρτης, ένα φύλλο πορείας, μια οδός που υποτίθεται ότι πρέπει να ακολουθηθεί και μετά βλέπουμε όταν υπάρξουν απρόπτα. πολλά μπορούν να προετοιμαστούν. το ξέρω ότι πολλές φορές δεν είναι ευχάριστα αυτά τα πράγματα, αλλά ε, η πλήρης διαφάνεια είναι ε, πάρα πολύ σημαντική. Όταν οι πελάτες δεν συμμετέχουν, δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι ε, και όταν τα στοιχεία ενεργητικού τους είναι αντικείμενο ανάκαμψης, αναδιάταξης για να μην πω εξυγίανσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τι τους περιμένει. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανισορροπία Ε, σε σχέση με τους πελάτες, διακριτική μεταχείριση εις βάρος τους, ε, σε σχέση με τους αντισυμβαλόμενους κτλ. Και ε, συμφωνώ με τον Φιλίπ, οποιαδήποτε ε, παρέκκληση από τους βασικούς κανόνες θα πρέπει να έχει μια επιβάρηση. Αλλά ποιος θα πληρώνει ε, και ε, τις πταίει. Τώρα μερικοί μπορεί να είναι πιο υπέτειοι από κάποιους άλλους και άλλοι μπορεί να είναι πιο υπεύθυνοι από ορισμένου. Θα τα δούμε αυτά και θα τα ορίσουμε ξεκάθαρα. Θα συζητήσουμε πάρα πολύ αυτά τα trigger points, τα σημεία που δρομολογούν τις εξέλιξεις που πυροδοτούν. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Υπάρχουν κάποια θέματα που καλύπτονται. Θα συζητήσουμε και τις υπόλοιπες τροπολογίες. Και μόλις θα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά, αρχίζει γενομένης από την επόμενη εβδομάδα, θα μπορέσουμε να ε, ψηφίσουμε. Πότε λίγη προθεσμία, 17 Οκτωβρίου. Ωραία. Ελπίζω να κάνουμε την ίδια πρόοδο μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, όντως. 17 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε αν μπορούμε και μετά στην Ολομέλεια τον Νοέμβρη με το καλό. Και μάλιστα το συντομότερο, όσο πιο γρήγορα κάνουμε τις προτάσεις μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο πιο εύκολα θα τις λάβουν υπόψη και χαίρομαι που συμφωνείς με αυτό το δρόμο που προτείνω να υπάρχει μια ε, στοιχειώδης έτσι, προσανατολιστική κατεύθυνση. Ε, ε, πάμε λοιπόν στο σημείο 16, λογαριασμοί πληρωμών, εξέταση των τροπολογιών, εισηγητής είναι ο Γιώργεν Κλούτερ. Θα ήθελα να σας θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι συνδέεται βάσει του άρθρου 50 η Επιτροπή ΙΜΚΟ ε, για την πρόσβαση του κοινού σε βασικούς λογαριασμούς πληρωμών. Δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Δεν ξέρω αν παρευρίσκεται η συγγήτρια της ΣΥΜΚΟ, όχι ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, ε, συντάκτρια μάλλον είναι γνωμοδότησης, έχει κάνει τροπολογίες και στην ΕΚΟΝ. Ζητήσαμε να είναι προτεραιότητα στους συντονιστές και να ψηφιστεί γρήγορα η έκθεση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να περάσουμε σε μια διαπραγμάτευση και να ολοκληρώσουμε μέχρι τα τέλη της θητείας τη συζήτηση με το Συμβούλιο. Και θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Όταν άρχισε η συζήτηση για τις αρμοδιότητες το θέλαμε και τότε, αλλά μάλλον η δουλειά άρχισε πολύ πρόσφατα μετά τη διάσκεψη των Προέδρων και τώρα λένε ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε πριν τις 27-28 Νοεμβρίου παρακαλώ παρόλο που συνεδριάζουν αυτοί και 4 και 5 Νοεμβρίου. Πρέπει να σας πω ότι το χρονοδιάγραμμα ΙΜΚΟ είναι απαράδεκτο τέλη Νοεμβρίου. Μα είναι διατρανωμένη πολιτική βούληση να προχωρήσουμε γρήγορα. και η αρμοδιότητά τους είναι μια μικρή ουρίτσα σε ένα τεράστιο σκυλί που είναι αυτός ο φάκελος. Μπορούμε, άμα, θέλ, άμα δεν θέλουν, να προχωρήσουμε ε, και να ψηφίσουμε στις 14 Νοεμβρίου. Δεν ξέρω, αν μπορεί κάποιος από σας να επηρεάσει την Επιτροπή ΙΜΚΟ, θα τους τα πείτε. Παρακαλώ. να μην μπλοκαριστεί αυτό, να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της παρούς εντολής. Ο Γιώργεν Κλούτε. Ευχαριστώ Σάρον. Μάλιστα. Μας εντυπωσίασε ο αριθμός των τροπολογιών. 734 παρακαλώ. Τροπολογίες έχουν κάνει συνάδελφοι για τους λογαριασμούς πληρωμών. Θα πρέπει βέβαια να το σχετικοποιήσουμε γιατί πολλές τροπολογίες μοιάζουν μεταξύ τους για διάφορα σημεία. Μπορεί να εντυπωσιάζει ο αριθμός, αλλά επί της ουσίας είναι λιγότερες. Αυτό όμως είναι ένα σημάδι ότι η Επιτροπή μας λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό και ψάχνει και λύσεις που να λειτουργούν για όλους τους ενδιαφερομένους και για τις υπηρεσίες πληρωμών αλλά και για τους χρήστες, δηλαδή τους καταναλωτές αλλά και το λιανικό εμπόριο, δημόσια διοίκηση και άλλους πελάτες των τραπεζών. Και βέβαια οι λύσεις που θέλουμε εμείς να προτείνουμε θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό κατά την άποψή μου Είναι καλό που συμμετείχαν και άλλοι συνάδελφοι, εκτός από τους σχεδοσυγητές, ε, από διάφορα κράτη-μέλη, γιατί ξέρουν πώς έχει πραγματικότητα στην κάθε χώρα. Για τις πληρωμές, για τη συμμετοχή του κοινού, δεν θα πρέπει όλα να τα ε, ευθυγραμμίζουμε προς τα κάτω ή προς την ίδια κατεύθυνση και να τα σιβερώνουμε έτσι ώστε να είναι απαντού ομοιόμορφα. Υπάρχουν και ε, πολιτιστικές διαφορές. Ε, κάποιοι λαοί, κάποιες χώρες έχουν ε, περισσότερη συνήθεια να χρησιμοποιούν μετρητά και δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει ένα καταναλωτή Sony και καλά να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Δεν είναι οδηγία που υποχρεώνει τους πελάτες με το στανιό να ανοίξουν ένα λογαριασμό σε τράπεζα αλλά αυτοί που χρειάζονται και θέλουν λογαριασμό να έχουν και το δικαίωμα να ανοίγουν. Ε, θεωρώ παρόλα αυτά ότι στην Επιτροπή μας τρία είναι τα βασικά που θα πρέπει να μας καθοδηγούν και δεν θα πρέπει να ε, τα ε, ξεχνούμε. Πριν αφήσω το λόγο στους κοιόδης και στους συναδελφούς, να επαναλάβω αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Και οι μεμονωμένες τροπολογίες καταλάβατε ότι δεν μπορούν να εξεταστούν όλες ε, στις λεπτομέρειες. Πρώτον, η οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο βήμα ε, για μια εσωτερική αγορά των λογαριασμών πληρωμών. Σήμερα ε, είναι κατακαιρματισμένα αυτά και δεν υπάρχει πρόοδος. Θα πρέπει να βοηθήσουμε να μεταξελιχθεί, να ξεπεραστεί αυτός ο κατακαιρματισμός και η πολυδιάσπαση ελευθερή κυκλοφορία εργαζομένων, ε, άρα δεν θα πρέπει να είναι άθλος να ανοίξει στην Ιταλία ή στην Αγγλία ε, ένα λογαριασμό ή να κλείσει το δικό σου λογαριασμό στη χώρα σου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερες δυσκολίες ε, να ανοίξουν λογαριασμό δεν είναι μόνο υπερχρεωμένοι αλλά και άστεγοι και άνθρωποι που ζητούν δουλειά, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι που θέλουν να πάνε σε μια άλλη χώρα, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και φοιτητέ. Έχουν συχνά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη τις ανάγκες και αυτών των πολιτών και εμείς ως βουλευτές δεν θα πρέπει να τον αμφισβητούμε καταρχήν, λέω εγώ. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Θα πρέπει να είμαστε στραμμένοι προς τα ευρώ αν θέλουμε ε, ε, η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι κατευθυντήρια νήμα και γραμμή και ερμός δεν μπορούμε να δηλώσουμε ικανοποιημένοι. Σε, αν κοιτάξτε τι ε, χρεώνουν οι τράπεζες για ένα προλογαριασμό στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία, δεν ξέρω αν φταίει μόνο ο πολιτισμός και οι συνήθειες κάθε χώρας. Τα υπερβολικά έξοδα μπορεί να είναι αποδοτικά για τις τράπεζες, αλλά για την οικονομία ε, είναι φραγμή. Στη συνέχεια, ανταγωνισμός όσο είναι ακριβή και επικίνδυνη και ε, ε, ρίσκο αυτή η διαδικασία, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Ε, σε μια αγορά ελεύθερη και οικονομία της αγοράς θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία οι καταναλωτές να αλλάζουν και τράπεζα. Και από πλευράς των τραπεζών, αλλά ε, στο ΕΛΚ, στο ECR και EFT δεν θέλουν να διευκολύνουν την ε, διασυνοριακή αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού και τράπεζας. Εγώ, άμα θέλετε, να συζητήσουμε και τα προβλήματα και τα εμπόδια, τα συγκεκριμένα που υπάρχουν, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, χώρες που δεν έχουν το ίδιο νόμισμα. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε καινοτόμοι και φιλική προς τους καταναλωτές που είναι και 500 εκατομμύρια στην Ένωση χρειάζεται ε, μια ρύθμιση ε, ε, για να προχωρήσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας τους καταναλωτές και όχι τα μικρό συμφέροντα των διαφόρων κρατών μέλων. Η έκθεση πρωτοβουλίας ε, έγινε δεκτή και στην Επιτροπή μας με μεγάλη πλειοψηφία που ζητάει όσο γίνεται πιο εύκολη πρόσβαση σε ένα λογαριασμό πληρωμών με τη λογική ότι ε, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται όταν λέτε ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές μόνο εφόσον έχει εγκριθεί από μια τράπεζα ε, το άνοιγμα ενός λογαριασμού. Δηλαδή τι, οι τράπεζες θα, θα το ε, ε, αποφασίζουν αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το δικαίωμα να ανοίγει λογαριασμό, όχι το δικαίωμα να σε πετάει έξω μια τράπεζα, γιατί ορισμένοι αυτό προτείνουν, πώς μπορούμε να δώσουμε παράθυρα και παραθυράκια και δυνατότητες στις τράπεζες, ε, για να απορρίπτουν ε, κάποιες συμπεριφορές ας πούμε και κάποιες τακτικές ε, των καταναλωτών. Θέλω να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ξεκάθαρα αυτό το τομέα και τον έχει περιορίσει πάρα πολύ και τον έχει στενέψει πολύ γιατί η συμπεριφορά είναι κάτι αφηρημένο, κάτι υποκειμενικό. Τι θα πει ανάρμοστη συμπεριφορά, απαράδεκτη συμπεριφορά, ε, εχθρική συμπεριφορά. Αυτό ποιο το αξιολογεί η τράπεζα. Και επίση ε, θέλω να πιστήσω την προσοχή σας και ε, στο εξή. Υπάρχουν και εγκληματικέ ενέργειες. Βλέπε ξέπλυμα χρήματος ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε. Προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτό. Αλλά πρόσφατα είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπου τραπεζών από τη Γερμανία και μας είπαν ότι τελικά το ξέπλυμα μόνο εκ των υστέρων το βλέπεις και ε, προχωράς σε νομικά βήματα. Εξάλλου, ε, ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε, η πελατεία μας για να το πω έτσι, δεν ξεπλένει χρήματα. Το ξέπλυμα υπάρχει από πάντα. Δεν θα γίνει τώρα με αυτούς τους λογαριασμού. Όταν δημιουργεί κάποιος ένα νέο εργαλείο, βέβαια υπάρχει πάντα έδαφος και για ε, καταχρήσει, αλλά δεν μπορούμε με υπερβολικές ε, ε, ε δυσκολίε και υπερβολικούς ελέγχους να προχωρήσουμε. Υπάρχει και το θέμα της υπόνοιας. Ωραία, γιατί ποιον θα υποπτευτώ εγώ για ξέπλυμα. Αυτό είναι θέμα των διοκτικών αρχών. Εισαγγελέα και αστυνομία επεμβαίνουν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις κλείνουν και τους λογαριασμούς. Αυτό δεν είναι θέμα της τράπεζας, είναι θέμα των διοκτικών αρχών. Είναι του ποινικού δικαίου. Δεν θα αποφασίσει μια τράπεζα ε, τι λογαριασμό θα μπλοκάρει και τι λογαριασμό θα κλείσει. Αυτό το θέμα της υποψίας ή της υπόνοιας είναι περίπλοκο. Δεν μπορεί να είναι στη διακριτική ευχαίρεια της τράπεζας. Αλλιώς τους ανοίγουμε κάποιες θύρες για δράση σε ε, τομέα που δεν είναι καθόλου φιλικός προς τους πελάτες. Αυτά. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Uh, Πολύ σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ακούσουμε τους κοιόδης. Ελκ, Λάγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θυμίσω λίγο ε, την ε, αιτιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι κοινωνική πολιτική, είναι εσωτερική αγορά. Για την κοινωνική πολιτική, σύμφωνα με τη συνθήκη, είναι θέμα επικουρικό για μας. Δεν έχουμε την κύρια αρμοδιότητα. Τι λοιπόν έχει σχέση με την εσωτερική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι υπάρχουν 58 εκατομμύρια 9% του πληθυσμού χωρίς τραπεζικό λογαριασμό και από αυτούς η μισή τα 25 εκατομμύρια θα ήθελαν να έχουν αλλά δεν τους ανοίγουν. Ε, την τελευταία πενταετία 16% των καταναλωτών έχουν αλλάξει τράπεζα, λογαριασμό. Άρα, ποια είναι η ανάγκη στη Βόρεια Ευρώπη μηδενική. Ε, έχουμε πλήρη κάλυψη, είμαστε εντάξει από βορρά προς νότο αφορά κυρίως αυτό δύο τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Αυτές είναι οι δύο λογοχώρες ε, όπου είναι μάλλον χαμηλή ε, η ε, λογαριασμοί σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό για το πώς έχει η κατάσταση τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα κράτη-μέλη, οδηγία είναι, οδηγία, και καλό είναι που είναι οδηγία γιατί θέλουμε να το ρυθμίσουμε, προτείνει τα κράτη-μέλη να δημοσιεύουν ένα κατάλογο με τράπεζες που ε, δίνουν τη δυνατότητα ενός βασικού λογαριασμού πληρωμών με ορισμένες ειδικέ λειτουργίες κτλ. και αποδείξεις. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό για τις πληρωμέ, το άλλο είναι να αλλάξει λογαριασμό και το τρίτο είναι ενιαία και διαφανή τέλη. Ωραία, αυτά είναι τα τρία. Άνοιγμα λογαριασμού. Αυτές είναι οι ειδικέ μου τροπολογίε και των συναδέλφων του ΕΛΚ. Δεν είναι αυτό που προτείνει ο κύριος Κλούτε σε κάθε κράτος μέλος να μπορεί ο καθένας να ανοίγει λογαριασμό και αυτό λέω και εγώ στην τροπολογία μου, ο καθένας το κράτος που μένει ή που έχει σχέσεις με τη χώρα. Δεν αρκεί ε, να πάω διακοπές στην Ισπανία, αλλά να σπουδάζω εκεί, να έχω ένα εξοχικό, εν πάση περιπτώσει, ε, να έχω κάποιους δεσμούς με τη χώρα. Ορίστε, αν είμαι φοιτητή εκεί, αν έχω τη δευτερεύουσα κατοικία μου, την εξοχική μου κατοικία. Όχι πήγα διακοπέ στην Ισπανία να ανοίξω ένα λογαριασμό. Αυτέ οι προποθέσει θα πρέπει να ορίζονται. Δεύτερον, προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει μεγάλο νόημα να πούμε ότι θα κάνουμε μια λίστα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τουλάχιστον 20 τράπεζες που προσφέρουν τέτοιο λογαριασμό βασικό πληρωμό. Κατά τη δική μου άποψη θα μπορούσαμε να υποχρεώσουμε κάθε τράπεζα να προτείνει ένα τέτοιο βασικό λογαριασμό πληρωμών. Κάθε τράπεζα. Έτσι. Αν περιορίζεται ε, σε πολίτες της Ένωσης που έχουν σχέση με τη χώρα. Είναι ε, ε, πολίτες της χώρας, έχουν την κύρια κατοικία, τη δευτερεύουσα, εργάζονται ή σπουδάζουν ένας τέτοιος βασικός λογαριασμός θα πρέπει να ορίζεται τι λειτουργίες έχει και τι προσφέρει και εδώ συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει μάλλον να είναι περιορισμένες οι λειτουργίες αλλά εάν κάθε τράπεζα προσφέρει ένα λογαριασμό ε, τότε ε, είναι πιο εύκολο να λυθεί το θέμα της διαφάνειας και του ανταγωνισμού. Το επόμενο θέμα, αλλαγή λογαριασμού. Γίνονται προτάσεις ότι έχει το δικαίωμα σε ένα λογαριασμό πληρωμών κτλ. Και, τα λοιπά, και όταν ε, τον καταγγέλεις και αλλάζεις τα ξεπλήματα χρήματος και όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε. αλλά γενικά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει μαζί με τα ξερά να κάψουμε και τα χλωρά, αλλά να αναγκαστούν οι τράπεζε να κάνουν τη δουλειά του, οι οποίε τα έχουν στυλώσει, γιατί λένε είναι πολύ ακριβά αυτά τα πράγματα, αλλιώ θα το προσφέραμε. Ε, αυτό το επιχείρημα δεν ευσταθεί. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι ελάχιστε προποθέσει, ούτε χρειάζονται τίποτα σπουδαίες εξίσου ερώτηση πράξη που θα βγάλουν ένα γραφικό τέρα, αλλά μπορούμε στα κράτη-μέλη να τα αφήσουμε σε μια οδηγία το πώ θα το διαμορφώσουν, εφόσον τηρούνται οι βασικέ προποθέσει. Και αυτή είναι η βασική προσέγγιση και γενική προσέγγιση που εγώ πρεσβεύω. Εντάξει, δεν έχω κάνει όλες τις τροπολογίες έτσι προς αυτή την κατεύθυνση, το έχουν κάνει άλλοι συνάδελφοι. Αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όμως προς την κατεύθυνση αυτή, πιστεύω ότι έχουμε μια λογική βάση για να προχωρήσουμε και να μην είναι στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών από το 2011 στην αυτοϋποχρέωση, αλλά σε μια διανόμου υποχρέωση. Αυτή είναι για μένα η σωστή οδός Βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις και έκτακτες περιστάσεις. Θα τα συζητήσουμε αυτά μεμονωμένα. Δεν θέλω να το πράξω εδώ και τώρα. Παράδειγμα, Όταν συμμετέχει κανείς σε μια συνεταιριστική τράπεζα, εδώ και καιρό εγώ συμμετέχω σε μια τέτοια ε, συνεταιριστική μετοχική τράπεζα, Raiffeisen, και μπορείς να ανοίξεις ε, λογαριασμό ή σε μέλος. Υπάρχουν τέτοια ταμιευτήρια στη Γερμανία που παρέχουν στα μέλη τους ε, τη δυνατότητα να ανοίξουν λογαριασμό. Ε, με κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Γι' αυτό έχω κάνει και την τροπολογία. Μια στιγμή να βρω τον αριθμό γιατί δεν τη θυμάμαι. 169 που λέγει ακριβώς ποιες είναι οι δυνατότητες, πακέτα, τραπεζικούς λογαριασμούς με προϊόντα κτλ. κτλ. Αλλά ε, και η συμμετοχή σύμφωνη με το καταστατικό απόκτηση της ιδιότητας μέλους συνεταιρισμού θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή σε λόγο επιμέρους διάταξης. Είναι 169 τροπολογία. Εμείς είμαστε υπέρ των καταναλωτών, δεν θέλουμε να διαστραβλώσουμε ε, τον ε, ανταγωνισμό. Εμένα δεν με νοιάζει να μπω στην ουσία του ανταγωνισμού και στη δομή του. Θέλω να υπάρχει μια βασική υπηρεσία προσφορά για τους καταναλωτές, όπως το ζητούν και σωστά πολλές οργανώσεις καταναλωτών, αλλά να μην κάψουμε, είπαμε, τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Και να μην μπορεί ο κάθε καταναλωτής να ανοίγει ένα λογαριασμό σε 28 κράτη-μέλη. αλλά να μπορεί να πληρώνει τους λογαριασμούς, τη ΔΕΗ, το νερό, ξέρω εγώ και τα λοιπά, από ένα βασικό λογαριασμό. Θα συζητήσουμε τι θα προσφέρει αυτός ο λογαριασμός, αλλά να είμαστε ανοιχτοί και να αναλύσουμε ότι αφορά κυρίως δύο κράτη-μέλη και μια υποψήφια χώρα ενδεχομένω που δεν έχει μπει ακόμα και λέγεται Τουρκία. Καλά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι του παρόντος, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε ένα λογικό συμβιβασμό πριν το τέλος της θητείας, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ελάχιστη ρύθμιση που να βοηθάει και τους ενδιαφερομένους χωρίς να δημιουργεί νέα γράφη ή οκρατία. Σας ευχαριστώ. Ε, thank Ευχαριστούμε. Λούτφιξον, σοσιαλιστής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν βλέπω αυτές τις τροπολογίες, ε, παίρνω πάρα ε, βλέπω πολλά υποσχόμενες ε, τάσεις. Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε πολύ καλές ιδέες σε σχέση με την αναβάθμιση της αρχής πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από τροπολογίες. Θα αρχίσει σύντομα η συζήτηση για τις τροπολογίες και προσβλέπω στην επικοδομητική συνεργασία που θα έχουμε. Ταυτόχρονα βλέπω τουλάχιστον τρεις βασικές ανησυχητικές τάσεις. Πρώτα απ' όλα από την άποψη των καταναλωτών. Ε, δεν υπάρχει τίποτα στις τροπολογίες, δεν είναι καλό αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι επικρατούν τα συμφέροντα των παρόχων υπηρεσιών και όχι των καταναλωτών. Ε, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πολλά και διάφορα εμπόδια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επανέλθουμε στη χρησιμότητα αυτής της πρότασης. πιο συγκεκριμένα να νομοθετήσουμε προς συμφέρον των καταναλωτών και όσο απλούστερα είναι τα πράγματα τόσο το καλύτερο. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος, η σημασία των καταναλωτών. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την ποιότητα του νομοθετήματος. Έτσι θα βελτιωθεί η κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ο ανταγωνισμός ε, θα ε, αυξηθεί ανάμεσα στις τράπεζες και θα μειωθούν οι οικονομικές ε, απώλειες. Αλλά πρέπει στο κέντρο, στον πυρήνα να είναι ο καταναλωτής για να συμβούν όλα αυτά. Επίσης, ε, είναι πάρα πολύ περίεργο που είναι κοντόφθαλμη και εθνική προοπτική υπό την οποία εξετάζουν κάποιοι το θέμα. Κάποιες ε, τροπολογίες ε, επικεντρώνονται μόνο στην, στην αποτροπή των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, ενώ υποτίθεται ότι προωθούν την ενιαία αγορά. Εγώ, το δικό μου εφαλτήριο είναι εντελώς διαφορετικό όταν εξετάζω το θέμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, να επιδιώξουμε, να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή κινητικότητα, Έχει το αντίθετο. Η τυποποίηση τώρα της ε, ορολογίας ε, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν νομίζω να είναι τόσο περίπλοκο πια αλλά θα έχει πολλά και σημαντικά ωφέλη για τη διασυνοριακή κινητικότητα. Συντρέχουν πολλοί λόγοι για να απόσχουμε από μια τέτοια στενή θεώρηση των πραγμάτων για να μην έχουμε μια χειρότερη κατάσταση σε ένα-δύο χρόνια στην Ευρώπη, να έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Ε, το σύστημα ΣΕΠΑ ε, ε, λειτουργεί καλά και Φυσικά, εντάξει, εξυπακούεται ότι υπάρχουν και επιπλοκές, αλλά νομίζω ότι με λίγη μικρή προσπάθεια μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πιο ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική αγορά και να μην περιοριζόμαστε στους, στις στενές εθνικές υποδομές. Έτσι θα καρκινοβατούμε αντί να πρόδευουμε. Επίσης ε, πρέπει να επιδιώξουμε τη μείωση των τελών για τις βασικές τραπεζικές ε, υπηρεσίες. Ο στόχος θα πρέπει να είναι όλοι, όλοι οι πελάτες να μπορούν να ανοίξουν και να έχουν αυτόν τον βασικό τραπέζικο λογαριασμό. Δεν μπορεί να αποκλείεται κάποιος επειδή και μόνο είναι ψηλά τα τραπεζικά τέλη. Το πρότυπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε γενικέ γραμμές είναι καλό, αλλά ξαναλέω πρέπει να ενισχυθεί σε ορισμένα σημεία, γιατί η διαφάνεια για τι τιμέ, γιατί αυτό συνδέεται με τους λογαριασμούς πληρωμών, διότι Ε, διότι ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί για ε, ε, μηνιαίες πληρωμές εφάπαξ ποσών. τώρα, σε σχέση με τις πληρωμές ε, για να βελτιωθεί η κατάσταση για τους ε, πελάτες. Ε, θα ήταν απλούστερο ένα διασυνοριακό σύστημα, αλλά οι αρχές θα πρέπει να είναι αντικειμενικές και κυρίως να επικρατήσει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη ορατότητα. Ε, τα κράτη-μέλη φυσικά το θέλουν μπορούν να θεσπίσουν ευνοϊκότερα για τους πελάτες συστήματα αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο πρότυπο και κάποια χώρα που θέλει να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να διευκολύνει τη ζωή των καταναλωτών θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να το κάνουν. Όταν μιλάμε για ένα λογαριασμό πληρωμών βασικών τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι καθολική ισχύωση διατάξεις. Ε, όλοι οι πάροχοι που προσφέρουν αυτή την υπηρεσία του βασικού τραπεζικού λογαριασμού ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ε, και ένα βασικό προσβάσιμο τέλος για αυτούς τους λογαριασμούς διότι προκύπτει και ένα Τίγμα αν θέλετε, αν υπάρχει μόνο ένας τραπεζικός οργανισμός που προσφέρει τέτοιου είδους λογαριασμούς και είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής να αποταθεί σε εκείνον. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τέτοιους μονοπόλια. Και να θεσπίσουμε ένα καθολικό δικαίωμα πρόσβασης ε, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και με άλλες κοινωνικές πολιτικές που έχουμε έτσι ε, ούτως ή άλλω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στις κατηγορίες των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι τράπεζε. αυτοί οι λογαριασμοί θα έχουν ναι, το χαμηλότερο δυνατό, το βασικό τέλος. Ε, οι καταναλωτές ε, δεν μπορεί να χρειάζεται να καταβάλουν υψηλό τέλο για τόσο βασικές υπηρεσίες. Τις επόμενες εβδομάδες ε, θα έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις ε, και είναι σημαντικό το νομοθέτημα για τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους παρόχους, στην ολοκλήρωση νέας αγοράς και για το σύνολο των καταναλωτών. Καταναλωτές που σήμερα δυσκολεύονται με ένα λογικό τέλος να έχουν πρόσβαση σε ένα βασικό τραπεζικό λογαριασμό είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχίσει και σε αυτό έγινε και μια πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Πολύ σας ευχαριστούμε, ε, λέει η Πρόεδρος ε, Φιλίπ Ντεμπάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από πλευρά φιλελευθέρων πρέπει να πω ότι συμφωνούμε και υποστηρίζουμε σε μεγάλες γραμμές την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι μόνο λίγες οι χώρες μέλη έχουν προβλήματα. Δεν είναι μόνο η Ρουμανία και η Βουλγαρία ε, που έχουν ε, μια κουλτούρα ε, χρησιμοποίησης μετρητών και είναι πιο δύσκολο να ανοίξει κανείς λογαριασμό ή να αλλάξει. Όχι, το αντίθετο, τις τελευταίες εβδομάδες είδα κάποιους όχι μόνο ε, στην ε, Ισπανία και στην Ιταλία, αλλά κάποιοι εργαζόμενοι στη Γερμανία που ζουν σε άλλες χώρες έχουν δυσκολία να ανοίξουν ένα λογαριασμό. Δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε στη μοίρα τους. Είναι καλή η πρόταση, αλλά ε, ε, και είναι δύο πράγματα. Είναι η κοινωνική συμπεριλήψη και η οικονομική. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, θέλει προσοχή και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ευαισθησίες και τις πρακτικές που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Γι' αυτό εδώ θέλω να ζητήσω μια στοιχειώδη επικορικότητα και να πούμε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι κοιτάξτε θέλουμε να έχουν ίση μεταχείριση οι πολίτες παντού στην Ευρώπη αλλά κάθε κράτος μόνο του να ε, στείνει το σύστημά του. Δεν μπορεί όλε οι τράπεζε να υποχρεώνονται ορισμένες τράπεζες ε, και να έχουν μια αντισταθμιστική ωφέλεια ή ακόμα και εθνικές τράπεζες ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει δυνατότητα ίσης μεταχείρισης ε, να πιστούν όλα τα κράτη-μέλη και δια της βίας ενδεχομένως να στήσουν ένα τέτοιο σύστημα. Και αυτό ακριβώς είναι μια οικονομική και κοινωνική συμπεριλήψη, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κριτήρια. Παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει μια διασύνθεση, μια σχέση ακριβώς με τη χώρα στην οποία ζητάς. Μα μου φαίνεται λογικό και για τον ε, οποιοδήποτε λογαριασμό για να καταπολεμηθούν φαινόμενα όπως είναι η απάτη και τέτοια. Επίσης, να είναι ένας βασικός λογαριασμός πληρωμών για να υπάρχουν εμβάσματα, πληρωμές και ε, να μπορεί κανείς να ε, κάνει ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό, από το ATM ας πούμε αυτά. Ε, επίσης η πρόταση έχει να κάνει και πολύ με την εσωτερική αγορά. Και εδώ σκέφτομαι κυρίως το πώς ε, μπορεί κανείς να μεταφέρει ένα λογαριασμό από μια χώρα σε άλλη. Και ε, θα ήταν σημαντικό βήμα για την κινητικότητα φοιτητών, εργατών και άλλων εντός της εσωτερικής αγοράς και έχω κάνει και τροπολογίες για δύο φάσεις και δύο στάδια. Πρώτον, το σύστημα ΣΕΠΑ που είχαμε και πριν από λίγα χρόνια προτείνει θα πρέπει να αναπτυχθεί, έχει ε, τεθεί σε λειτουργία, αλλά αν κάποιο κράτος μέλος ή μια τράπεζα δεν είναι σε θέση ή δεν θέλουν πρόθεσμα να υιοθετήσουν αυτό το σύστημα, τότε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία για διασυνοριακή αλλαγή η μεταφορά τραπεζικού λογαριασμού. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ε, γιατί ενδιαφέρονται πολλοί οι άνθρωποι. Επίσης όταν κάποιος θέλει να αλλάξει λογαριασμό ε, και διασυνοριακά ε, χρειάζεται μια στοιχειώδης διαφάνεια και συγκρισιμότητα και είναι και προς το συμφέρον του καταναλωτού και να κερδίσει μόνο έχει αν εναρμονίσουμε όχι μόνο την ορολογία αλλά και τη διαφάνεια. Και εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε και να είμαστε συνεπείς, όχι μέχρι τελευταίας και αρέας και κόμματος και τελείας, να έχουμε μια οδηγία με γενικές αρχές ε, που μπορεί να είναι συγκεκριμένες αλλά και συνεκτικές για να μην υπερφορτώσουμε τη βάρκα και την γραφειοκρατία, να υπάρχει δυνατότητα ε, λειτουργίας του συστήματος. Με δύο λόγια είναι σημαντική η πρόταση. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση. Δεν έχει να κάνει με ένα-δύο σημερινά κράτη-μέλη, ένα μελλοντικό κράτος. Είναι πιο βαθύ το ζήτημα και πραγματικά ελπίζω ε, και προσβλέπω και στις επόμενες συζητήσεις με τους ε, ε, εισηγητές να τα βρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σβέν Γκίγκολτ από τους Πρασίνους. Εδώ λέει πράσινη, πριν τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, δεν ξέρουμε ποια σειρά είναι. Uh, uh, My impression is that uh, always if Kamal and me we are shadowing, he always. Ε, έχω την εντύπωση ότι ο Καμάλ πάντοτε μιλάει μετά από μένα, δεν ξέρω γιατί, τέλο πάντων. Ε, Βέρνερ, από την περασμένη Κυριακή το έχετε πάρει τα πάνω σας βλέπω, δεν κρατιέστε. Από πριν, ναι, ναι, το πιστεύω και πριν έτσι ήσουνα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ ισχυρή η υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων, διότι ανελήφθηκε κοινή πρωτοβουλία από το Κοινοβούλιο και έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και κατόπιν πρόταση Εμένα, εγώ ασχολούμαι με την προϊούσα διαδικασία. Δεν είμαι σίγουρος ότι ε, το επεξεργάζεται το ζήτημα το Συμβούλιο και αν έχουμε χρόνο, καλό θα ήταν να ακούσουμε κανέναν εκπρόσωπο από την Επιτροπή και κυρίως από το Συμβούλιο να δούμε εκείνοι σε ποιο σημείο βρίσκονται. Διότι είναι μάλλον άχρηστο αν εκείνοι δεν εργάζονται για αυτό το ζήτημα, εμείς δεν πρόκειται να έχουμε ε, απτά αποτελέσματα. Αφήστε που πολλά ζητήματα σχετίζονται με τους καταναλωτές. Γιατί είμαστε τόσο επιλεκτικοί, είναι τόσο επιλεκτικοί στο Συμβούλιο και ε, ασχολούνται με τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν ε, επιλεκτικά. Είναι ε, ε επίσης ζήτημα νομικής βάσης. Και τώρα θα μιλήσω στα γερμανικά για να με ακούει και να καταλαβαίνει καλά ο κύριος ε, Λάγκεν. Όχι κανένα πρόβλημα μιλήσω γερμανικά. Χαίρομαι που ε, επανήλθαμε σε μια κοινή βάση. Είδα σε ένα ανακοινωθέν τύπου ότι ήσασταν είχατε πολλούς ενδιασμούς, ήσασταν μάλλον αντίθετος γιατί ισχυριζόσασταν ότι για λόγους επικουρικότητας δεν πρέπει να επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έγινε τώρα και επαναχωρήσατε. Εφόσον μιλάμε για την πρόσβαση στην ενιαία αγορά αφενός και αφετέρου για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ε, δεν αλληλοξιδετερώνονται αυτά. Έχουμε το άρθρο 114 ε, που αυτό αφορά και στην ενιαία αγορά και στην υψηλή προστασία των καταναλωτών. Ιδού λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτό. Τι γίνεται τώρα. Ε, υπάρχουν πολλά σημεία στην πρόταση όπου το υψηλό επίπεδο προστασίας αμφισβητείται. Ε, είναι το νήμα της Αριάδνης ε, που διατρέχει ολόκληρο το, το κείμενο. Επίσης έχουμε το άρθρο 3, δηλαδή σε ποιο μέτρο θα πρέπει τελικά τα μέτρα που θα αναλυθούν να είναι διαφανή πέρα από την το βασικό λογαριασμό. Μιλάμε και για την αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού. Ε, συνάδελφοι από το ΕΛΚ, από το, τους Φιλελευθέρους και το ECR κάνουν τροπολογίες που αποδυναμώνουν διατάξεις περί διαφάνειας. Το θέμα των τραπεζικών τελών, άρθρο 5. Υπάρχουν και προτάσεις για τη μείωση, ε, για την κατανομή στο άρθρο 7 κάτι που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση για οι κριτικές ιστοσελίδες να έχουν ως μόνο γνώμονα της σύγκρισης την τιμή. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ε, έολο. Δηλαδή συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Μια τραπεζά που προσφέρει μία μόνο η υπηρεσία είναι ε, στην ίδια μοίρα με μια τράπεζα που έχει πάρα πολλά υποκαταστήματα, ATM και τέτοια και μια σειρά άλλων υπηρεσιών. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια, όχι μόνο τα τραπεζικά τέλη και πόσο κοστίζει να ανοίξει ένα λογαριασμό, γιατί ε, ο ανταγωνισμός θα είναι προς τα κάτω ε, για τον πιο συμφέροντα και τον πιο φτηνό που δεν με ενδιαφέρει. Ε, αυτή η προσέγγιση και δεν είναι σωστή. Επίσης, ε, ποιοι θα πρέπει να προσφέρουν όλες αυτές τις τραπεζικές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει «Α, ας είναι και μια τράπεζα ένα χώρα μέλος». Μα για μένα αυτό επίσης τρευλώνει τον ε, γιατί αν τους δύσκολους πελάτες τους αφήνω σε μία μόνη τράπεζα και όλοι οι άλλοι απαλλάσσονται, ε, τότε πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και στη Γερμανία σε πολλά κρατήδια υπάρχει υποχρέωση για τα ταμιευτήρια, η Sparkassen. Γι' αυτό υποστηρίζω και τη γραμμή Langen που λέει όλοι να προσφέρουν την υπηρεσία γιατί η κοινωνική ευθύνη ε, αφορά όλους και το κόστος αυτό να το επομίζονται όλοι για το πώς θα εντάξουμε στην κοινωνία κάποιες δύσκολες ομάδες πολιτών και όχι ορισμένοι μόνο. Ε, παρακαλώ λοιπόν ε, όλες οι τράπεζες να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. Επίσης, ποιος θα έχει πρόσβαση και υποστηρίζω αυτό που είπε ο Φιλίπ Ντεμπάκερ. Δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, αλλά έχουμε τα προβλήματα αυτά ε, σε διασυνοριακούς εργαζομένους και στη Γερμανία πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει ως πρόσφυγες, de facto δεν έχουν αυτή την πρόσβαση. Και αυτή η έννοια του legal resident που έχει ε, χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ε, δηλαδή να είναι νόμιμα διαμένων, να είναι η βασική έδρα του στη χώρα, δεν είναι όλοι legal residents, παρόλα αυτά χρειάζονται τραπεζικό λογαριασμό για να λειτουργούν ως συμπολίτε και με την οικονομική έννοια του όρου. Μετά είναι το θέμα του ξεπλήματος του χρήματος. Γιούργεν, κλούτε, συμφωνούμε σχεδόν σε όλα. Αλλά εδώ έχω λίγο την αίσθηση ότι έχεις ε, απορροφήσει πολύ εδώ πέρα το φιλελευθερισμό. Και βέβαια υπάρχουν ε, ε, υποχρεώσεις ε, για το ξέπλυμα χρήματος και δεν είναι μόνο των διοκτικών αρχών εισαγγελίας και αστυνομίας. Παντού και δια νόμου μπορούν και οι τράπεζες να κάνουν έλεγχο ταυτότητας και παρακαλώ να το βάλεις και αυτό για τη διαφάνεια. Τώρα διαπληκτιζόμαστε για το πώς θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό σε πολλούς τομείς ακριβώς και θέλει μεγάλη προσοχή αυτό αυτή την ευθύνη να μην την ε, μεταφέρουμε μόνο στις διοκτικές αρχές, αλλά όταν κάποιος δραστηριοποιείται κάπου εμπορικά και οικονομικά, θα πρέπει παρακαλώ να υπόκειται και σε έλεγχο ε, και στα πιστοτικά ιδρύματα να υπόκειται και στην αστική ευθύνη. Βέβαια, ε, με όλα αυτά που συζητάμε έχει μικρή σχέση το θέμα και δεν θα πρέπει να βάζουμε επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται ε, για να υπεφεύγουν ε, όλοι ή κάποιοι και να αποποιούνται τις ευθύνες τους. Αυτά. Θα πρέπει το συντομότερο να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα για να μην βρίσκει δικαιολογίες ε, το Συμβούλιο και δεν ολοκληρωθεί στην παρούσα θητή αυτή η προσπάθεια. Οι συντονιστές το έχουν ξεκαθαρίσει το Συμβούλιο ότι θέλουν να γίνει τώρα. Θέλουν οι πολίτες και ένα σημάδι και ένα σύμβολο ότι ε, οι φορείς ε, των τραπεζών και της αγοράς δεν ενδιαφέρονται μόνο για τη σταθερότητα των τραπεζών και των τιμών αλλά και για τους συμπολίτε μας που είναι σε πιο αδύνατη θέση και κινδυνεύουν με κάποιους αποκλεισμούς. Αυτό είναι πιο σημαντικό από τις μικρές διαφορές που μπορεί να έχουμε σε μικρές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, Σάιεντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω ήδη καλύφθηκαν. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει συγκρισιμότητα των τελών. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφέρθηκε. Είναι το εξή. Κάποιο δανείζει 90 ευρώ σε κάποιον και του ζητάει να του δώσει πίσω 100 ευρώ. Ε, αυτό ε, σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι τεράστιο επιτόκιο, έτσι. 2.000% σε ορισμένους ε, χώρες ε, υπάρχουν διαφορετικές ε, νοοτροπίες σε σχέση με το ποια τέλη είναι αποδεκτά και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν. Χρειάζεται η λύση αυτή να γίνει σε εθνικό επίπεδο, όχι να αποφύγουμε το ευρωπαϊκό, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διαφορετικά συναλλακτικά ήθη σε κάθε κράτος. Συμφωνώ με τους συναδέλφους από το ΕΛΚ και από την ΑΛΤΕ για την αλλαγή τράπεζας. που η οποία αφορά περισσότερο την ε, επιλογή να αλλάξει κανείς τράπεζα εντός της χώρας του παρά να πάει από μια ε, χώρα στην άλλη. Ο στόχος μας στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν να δημιουργηθεί ένα σύστημα με το οποίο μπορεί κανείς να αλλάξει τράπεζα σχεδόν αμέσως. Και είναι ε, ζήτημα πληροφοριακών συστημάτων. Εγώ εργαζόμουν πριν από σχεδόν 20 χρόνια στον τομέα και ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει η μεταβολή αυτή μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο. Αλλά το ερώτημα αν υπάρχει ζήτηση. Εάν υπάρχει ζήτηση στο ε, μέλλον, νομίζω ότι αυτή θα εστιάζεται περισσότερο στο δικαίωμα του καταναλωτή να αλλάξει τράπεζα εντό της χώρας του και όχι από τη μια χώρα στην άλλη. Διαφορετικά, θα μπορούσε κανείς να καταχρηστεί το σύστημα και να δημιουργήσει λογαριασμούς 28 ε, κράτη-μέλη και αυτοί οι λογαριασμοί να μην είναι διασυνδεδεμένοι. Προφανώς δεν σας κατηγορώ κύριε Κλούτσε, ότι σκοπεύετε να κάνετε κάτι τέτοιο ή ότι σκοπεύετε να διευκολύνετε το ξέπλυμα, αλλά ε, για να μπορεί κάποιο να έχει δικαίωμα να ανοίξει ε, λογαριασμό σε μια χώρα θα πρέπει να έχει ένα σαφέ δεσμό με αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι εμεί ξεκινάμε από την αφιτερία τη ενιαία αγορά, τη κοινή αγορά. Ε, το, το τέλος ΣΕΠΑ, στο τελικά, είναι μηδαμινό. 9, από 9 λίρε το μειώσανε μάλιστα σε 4 ε, λίρες για διασυνοριακή συναλλαγή ΣΕΠΑ τη τραπεζά μου. Λοιπόν, πόσο πιο χαμηλά θα, θα, θα, θα φτάσει αυτό. Ίσως είναι ε, πιο εύλογο κάποιο να κάνει διασυνοριακές συναλλαγή ΣΕΠΑ παρά να ανοίξει ένα λογαριασμό στην χώρα. Υπάρχει κάτι που λείπει σε αυτή την συζήτηση ο πατέρας μου ήρθε το 50 στην ε, Αγγλία και θυμάμαι ότι πλήρωνε συνέχεια με μετρητά. Δεν τον ενδιαφέραν οι τράπεζε, δεν χρησιμοποιούσε πιστοτικέ κάρτε και τέτοια. Και το ερώτημα είναι γιατί θέλουμε να αποκλείσουμε εκείνου που θέλουν να χρησιμοποιούν μετρητά. Γιατί δηλαδή να του τιμωρούμε εκείνου που επιθυμούν να πληρώνουν με μετρητά και όχι να ανοίξουν λογαριασμό σε μια τράπεζα. Όταν ανοίγει ένα λογαριασμό μια ε, τράπεζα, ε, αναγκάζεσαι να πληρώνει κάποια τέλη, για παράδειγμα για τα εξτρέ και τα λοιπά, και αναγκάζεσαι να πληρώνει και να χρησιμοποιήσει αυτόν τον λογαριασμό. Γιατί λοιπόν να αποκλείουμε εκείνου του πολίτε οι οποίοι ε, και είναι ακριβώ εκείνοι που έρχονται από τι πιο μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδε, επιθυμούν να πληρώνουν με μεριτά. Αυτοί δεν θα πρέπει να τιμωρούνται ή να αποκλείονται. Απ' τη μία ασκούμε κριτική στις τράπεζες και συχνά ε, λέμε ότι οι υπηρεσίες του προς τους πελάτες πέφτουν και η εμπιστοσύνη προς αυτές χάνεται ταυτόχρονα μας ζητάμε από αυτές τις τράπεζες να ε, εξυπηρετούν τις μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες. Αυτό που θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε θα είναι περισσότερο ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών σε αυτόν τον τομέα. Και δεν το συζητάμε περισσότερο. Θα έπρεπε περισσότερο, για παράδειγμα, να αξιοποιήσουμε τι τεχνολογικέ λύσει. Στην Αφρική, για παράδειγμα, οι ε, πληρωμέ μέσω κινητού τηλεφώνου είναι πρωτοπόρη σε αυτό. Οι, οι, πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου δεν μπορούσαν να μειώσει το κόστος για τις τράπεζες. Είναι πιο φθηνή για εκείνες. Ε, Επίση οι προπληρωμένε κάρτε είναι μια λύση. Όταν χωρίς κανείς να έχει λογαριασμό μπορεί να έχει μια τέτοια κάρτα και να ε, προσθέτει όταν έχει χρήματα να προσθέτει ε, credits. Να αποθηκεύει, να αποταμιεύει τα χρήματά του σε αυτή την προπληρωμένη κάρτα και με αυτήν την προπληρωμένη κάρτα να πληρώνει τους λογαριασμούς του. Επομένως θα έπρεπε να προσπαθούμε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, όχι να τους δίνουμε όλο και περισσότερες εξουσίες και αρμοδιότητες και παρέμβαση με στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σέμπο δεν είναι εδώ, επομένω έχω ένα μεγάλο κατάλογο ομιλητών. Ας, λοιπόν, να σας αναφέρω τον κατάλογο των ομιλητών, έτσι ώστε να τον γνωρίζουμε όλοι. Myself, Peter Simon, Jean-Paul Gauges, Werner Langen has been waving as if he wants to come back in again, um, but, uh, uh, well, can't, you, you should have told Astrid. Anyway, um, Astrid. Astrid, έχετε το λόγο. Καλά, θα είμαι σύντομη, γιατί τα είπαν όλα οι προηγούμενοι, κυρίως ο διπλανός μου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του δεν νομίζω να βρεθεί και κανένας που να είναι κατά της έγκρισης τέτοιων προτύπων ε, και της κατοχήρωσης της πρόσβασης για όλους τους πολίτες σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Πολύ καλή είναι αυτή η ιδέα και την υποστηρίζω πλήρως. Βεβαίως είναι προς συμφέρον όλων να εφαρμόσει τα πρότυπα και ο τραπεζικός τομέας. Όμως προσοχή, ας μην υπερβάλλουμε διότι μπορεί να δυσχεράνουμε ή και να καταστήσουμε αδύνατο αυτό που εμείς κρίνουμε απαραίτητο. Ε, η πρόσβαση, λοιπόν, καθολική πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, γιατί μπορώ να το εκφράσω έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο στο κράτος διαμονής κάθε πολίτη. Αυτό μου φαίνεται προφανές. Δεν θα προβλέψετε ένα κανόνα που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να προσφέρουν τέτοιο λογαριασμό και να μπορεί ο πολίτης σε όλα τα κράτη-μέλη να ανοίξει ένα τέτοιο λογαριασμό. Δεν γίνονται αυτά. Είναι γελία θα έλεγα. Εντάξει να έχουμε την πρόσβαση σε μια βασική τραπεζική υπηρεσία και ο κ. Λάγκεν ή οποιοδήποτε, οποιοσδήποτε άλλος ε, απέφχεται την, ε, τη δυνατότητα ανήμως λογαριασμού σε 28 κράτη-μέλη. Αλλά όντως, όντως θα πρέπει να προβλέπετε αυτό μόνο για τους νομίμους διαμένοντες σε ένα κράτος. Αλλιώς δεν γίνεται στην πράξη και ξαναλέω ότι είναι και λίγο ανόητο και γελίο διότι συνεπάγεται αυτό τέλει που θα μετακυληθούν στους υπόλοιπους πελάτες της τράπεζας. Και συμφωνώ με τον Βέρναν δεν πρέπει να είναι μία μόνο η τράπεζα, ένα κράτος μέλος, διότι ποια φήμη θα έχει αυτή η τράπεζα. Μάλλον κακή. Θα είναι η τράπεζα των φτωχών, πώς θα τη λέμε. Είναι επιβλαβές. Όλες οι τράπεζες πρέπει να το κάνουν και δεν βλέπω και γιατί όχι. Αυτά που είπατε για τους ε, όσους διαμένουν στις μεθορίους. Εμείς έχουμε 160.000 τέτοιους. Για ένα συνολικό πληθυσμό 515.000 και τι, εργάζονται στο Λουξεμβούργο, εκεί πληρώνονται εκεί πληρώνουν τις φορές τους την κοινωνική ασφάλιση. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα και αν κάποιοι προβάλλουν αντιρρήσεις να μας το εξηγήσουν γιατί. Πού εσείς τους τα παίρνετε τώρα τα λεφτά. Ε, άμα έρθεις με μαύρα λεφτά δεν σου ανοίγει κανείς λογαριασμός να ξεπλύνεις. Γελάει ο κύριος Λάγκεν. <laughs> mais c'est vrai. Μα καλά αλήθεια είναι αυτά που λέω. Θα τα πω γερμανικά για να τα καταλάβεις. Εγώ θα επιθυμούσα όλες οι χώρες να είναι τόσο αυστηρές για τις καταθέσεις σαν το Λουξεμβούργο. Αυτό τώρα βγήκε, λέει ο κ. Λάγκεν, τώρα μας προέκυψε. Όχι. Και σταματήστε να διαδίδετε τέτοιες ανοησίες και βλακίες. Είναι πάρα πολύ αυστηροί οι λογαριασμοί στο Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ Άστριτ που με ανακάλεσε στην τάξη. Ε, μη μου λες τώρα τέτοια... Εγώ νομίζω είναι λογικό και απαραίτητο να διευκολύνουμε και τη μεταφορά των λογαριασμών από τη μία τράπεζα στην άλλη, γιατί ορισμένες φορές υπάρχουν κολλήματα, υπερβολικά πολλά κολλήματα, διότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να κρατάνε την πελατεία, αλλά και πάλι εδώ ε, θα πρέπει να σχεδιάσουμε τα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο, ε, είναι ε, ψευδέσεις ή το να πιστεύει κανείς ότι θα συμμορφωθούν τράπεζες σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο εύκολα όσο σε εθνικό επίπεδο. Όχι ότι θέλω να αναχαιτήσω αυτή τη γενική τάση των διασυνοριακών ε, αλλαγών ε, λογαριασμών, αλλά όταν ε, μιλάμε για τις απαιτήσει, ε, ας ξέρουμε και συνειδητοποιούμε ότι η ενιαία αγορά πόρο απέχει από την εσωτερική αγορά. Να πω στα γερμανικά κάτι στο συνάδελφο Γκίγκολτ, διότι είπε κάτι για τον κύριο Κλούτε. Θεωρεί ότι ο κύριος Κλούτε ε, έχει απορροφήσει ή τον έχει ρουφήξει ο φιλελευθερισμός. Πότε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο να σκεφτούν οι πράσινοι γιατί πήρατε λιγότερες ψήφους στη Γερμανία από ότι αριστερά, η Λίνκε. Okay, Astrid, you finished. <laughs> Astrid, τελείωσες. Τελείωσα. Right. Um, okay, we've got some coalition busting. Μάλιστα, σπάνε συνασπισμοί εδώ, γίνεται χαμός. Ε, κάθε. Ευχαριστώ, Σάρεν. Ε, ε, αυτά που είπε η κυρία Λούλινγκ για τη, μεταφορά των, τη δυνατότητα μεταφοράς ε, των λογαριασμών από τη μία χώρα στην άλλη και το ένα ίδρυμα στο άλλο. Κοιτάξτε, δεδομένης της νέας τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, ε, πιστεύω ότι είναι δυνατό, αν το επιλέξετε, να αλλάξετε τραπεζικό λογαριασμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει συμβεί αυτό παρότι ε, χρειάζονται θεωρητικά εννέα μέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο για να γίνει αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κάνει ε, αξιολόγηση κόστους ωφέλους για αυτό το ζήτημα της μεταφοράς γιατί σε τέσσερα-πέντε χρόνια θα την έχουμε την τεχνολογία πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Ε, παρότι σήμερα εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα για τους ε, λογαριασμούς ε, πληρωμών και ελπίζω να μην βαριέστε με αυτά που σας λέω, αλλά πρέπει να μοιραστώ μαζί σας κάποιες εμπειρίες που είχα. Παραδείγματο χάρη για τους παιδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ένα άλλο θέμα που πρέπει να διερευνηθεί και πιστεύω ότι είναι οι ευπαθέστεροι κατάλληλοι. Και επίσης όλοι όσοι φροντίζουν για το μέλλον του παιδιού τους. Ε, είναι, χωλένουμε ε, ως προς αυτή την υπηρεσία. Τέλος, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες ε, για την υποστήριξη των πιστοτικών ενώσεων, εγώ ανήκω στην τοπική ένωση και ναι, εντάξει, είναι, έχουν τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά παρόλα αυτά προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Ας μην υπονομεύσουμε το έργο τους. Ευχαριστούμε, Σάρων είτε ευχαριστώ πολύ για αυτό μου είπες. Τώρα κατάλαβα γιατί ο κύριος Ζέχοφερ απέκλεισε ε, συζητήσεις για σχηματισμό κυβέρνησης με τους πρασίνους, αλλά όχι με την αριστερά, τη Λίνκε. Ε, μάλλον αυτό που είπατε θα φταίει και εγώ αν ήμουν αριστερός ε, θα πρόσεχα πάρα πολύ μήπως είμαι το επόμενο θύμα αυτής της ιστορίας. Ναι. Έχω εγγραφεί και εγώ στο ε, κατάλογο γιατί έχω κάνει τροπολογίες. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή η ιδέα το να μπορεί δηλαδή κάποιο να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό ε, εκ των προτέρων σε μια χώρα πριν φτάσει. Δηλαδή να μπορεί να έχει ανοίξει το λογαριασμό. Ένα από του γιου μου χρειάστηκε να το κάνει το περασμένο Σάββατο γιατί έφυγε, πήγε να δουλέψει στην Ιρλανδία. Πολύ εκνευριστικό, πάρα πολύ να μην μπορεί να το κάνει αυτό εύκολα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αποδείξει ότι θα απασχολήσει εκεί και να υπάρχει μόνιμο σύνδεσμο με τη χώρα ή να αποδείξει ότι θα μένει εκεί. Τέλος πάντων, ένα ουσιαστικό σημείο συνδέσμου χρειάζεται για να ε, στοιχειοθετήσεις ότι πληρείς τι προποθέσει για την καταπολέμηση τη νομοποίηση των ε, εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. αλλά αυτό ισχύει και για του κανονικού λογαριασμού, όχι μόνο για του βασικού. Ε, τώρα για το αν θα είναι ένας ο πάροχος ή περισσότεροι. Ε, πρέπει να είναι τουλάχιστον αρκετά μεγάλος, ώστε όπου και να είστε στην επικράτεια του κράτους μέλους, ε, οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση. Δηλαδή, σε τι ωφελεί να ορίσουμε έναν ε, πάροχο, όπου όμως δύσκολα θα έχουν όλοι πρόσβαση, λόγω της τοποθεσίας. Εάν δεν επιδιώξουμε την ε, συνολική λύση, όλοι δηλαδή να υποχρεούνται να προσφέρουν τέτοιο λογαριασμό, ας έχουμε τουλάχιστον κριτήρια. Ε, τι συνιστά, τι, ε, από τι αποτελείται αυτή η επαρκή, σε βασική υπηρεσία. Υπάρχει και το θέμα της παιδείας των καταναλωτών. Πολύ ωραία να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμούς. Αλλά αλλά να ξέρουν και πώς να το χρησιμοποιούν. Ε, ξέρετε αυτές οι απάτες με τις επιταγές που οπισθογραφούνται και πάτε και ε, καταβάλλετε το ποσό στο όνομα κάποιου και αυτό γίνεται διασυνοριακά. Θυμάστε πόσο χρόνο μας πήρε για να σταματήσει αυτή η υπόθεση. Ποιο λέει σε κάποιους τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Είτε μιλάμε για επιταγές, είτε για τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε οποιαδήποτε άλλα εργαλεία ή σε ε, ένα περιβάλλον όπου δεν είναι κάτι συνηθισμένο να έχεις τραπεζικό λογαριασμό. Α πάρω και το προσωπικό μου παράδειγμα. Ε, η, μητέρα μου μου τα είπε τα περί τραπεζικών λογαριασμών και όχι η τραπεζά μου. Transparency and, ε, για τα τέλη, για την, τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις τράπεζες και τα λοιπά. Είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι για τα επιτρεπόμενα σε σχέση με αυτά που ακούσαμε και γιατί να μην κάνουμε ευρύτερε συγκρίσει με προϊόντα που προέρχονται από άλλους τομείς. Ε, όχι ότι θέλω να μπερδευτούμε τελείως, αλλά θα ήταν πρόβλημα να ορίσουμε τους ελάχιστους κανόνες. Ούτε θέλω να προσπαθήσουμε να απαγορεύσουμε το ε, κάποια είδη... Κα, κάποιους παρόχους, αν είναι από το δημόσιο ή από την ιδιωτικό τομέα, Ε, και για τις ιστοσελίδες αυτών των ιδρυμάτων ε, ε, εάν αποδειχθεί και ότι είναι παρικούς ποιότητας, ικανοποιητικής ποιότητας δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα τι γίνεται. Εάν αρχίζουμε να επανεξετάζουμε την ιδέα της ε, ε, άνευ χρέωσης τραπεζικής ε, υπηρεσίας. Τι σημαίνει αυτό δεν υπερβολικό άλλοι να πληρώνουν καταχρηστικά υψηλά τέλη όπως παραδείγματος χάρη μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν να πληρώσουν ούτως ή άλλως και θυμάστε όταν ασχολούμασταν με την οδηγία για τις πληρωμές στην προηγούμενη θητεία αυτό μας είχαν πει και μας είχαν πιστεί στην προσοχή μας και δεν είμαι σίγουρη ότι ε, το έχουμε φροντίσει αυτό και συνήθως ε, θύματα πέφτουν οι μικρομεσές γιατί τους μεταχειρίζονται σαν ιδιώτες ε, οι τράπεζες, κυρίως οι ιδιωτικές τράπεζες. Κάποιοι που ψήφισαν υπέρ των ιδιωτικών τραπεζών για τους ιδιώτες, ψήφισαν με την ιδιότητα μέλους ή συνεταίρου μικρομεσαίας επιχείρησης. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε πράγματα που επιχορηγούνται από άλλους ε, έμεσα κιόλα. Ε, πρόκειται για κοινοφελή υπηρεσία, είναι κάτι διαφορετικό έχουμε σε κάποια κράτη-μέλη εκτεταμένες διατάξεις για την αλλαγή λογαριασμού, αλλά δεν πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό. Ας μεγιστοποιήσουμε τις ε, διατάξεις. Αν ένα κράτος μέλος έχει ευνοϊκότερες διατάξεις, θα τις κρατήσει και ε, γιατί μπορεί να έχει επενδύσει σε αυτό το νέο σύστημα και τέλος ε, αυτό είναι οδηγία ούτως ή άλλως. Ε, άρα, αν χρειαστούν επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των μέτρων, τότε θέλω ένα άρθρο στο διατακτικό που να λέει ότι αυτή είναι η βασική απέτηση της ΕΚΟΝ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που ε, περιορίζεται όλος ιδιαίτερος σε αυτές τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λόγω του ρόλου των εθνικών εποπτικών αρχών όταν ελέγχουν το αν είναι ε, μία δραστηριότητα νομότυπη. Ωραία, Ζήμων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, δεν ξέρω τι είναι πιο παράλογο ε, να μας θεωρούν νεοφιλελευθέρους εμάς ή κάποιος να έχει 28 τραπεζικούς λογαριασμούς ε, σε 28 κράτη-μέλη. Ποιος μπορεί να είναι τόσο βλαμμένος και να πάει σε 28 χώρες να ανοίξει 28 λογαριασμούς. Τι είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα τέτοια πράγματα. Ξέπλυμα χρήματος με ένα βασικό λογαριασμό με ελάχιστες ε, υπηρεσίες. Δεν νομίζω να είναι οι απαταιώνες τόσο αδαείς και τόσο ηλίθιοι. Ε, και ε, τα είπα αυτά γιατί είχα μπει στον πειρασμό να μιλήσω κι εγώ για την ενδογερμανική συζήτηση. Δεν, δεν άντεξα. Λοιπόν, ε, είπαμε ότι ε, δεν θα πρέπει να περιορίζουμε τη συζήτηση. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια διεύρυνση, όπως είπε και ο συνάδελφος Λούτβιξον, για να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά και να φροντίσουμε ε, όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση. Και όχι μόνο αυτοί που έχουν την έδρα τους και την κατοικία τους σε κάποιο κράτος μέλος. Ούτε οι διασυνοριακοί υπάρχουν και άστεγοι. Πώς θα τους βοηθήσω ε, να φύγουν από αυτό το φαύλο κύκλο. Δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν τράπεζα, ε, ε, δεν έχουν διεύθυνση. Κάτι από όλα αυτά πρέπει να αποκτήσουν για να έρθουν και τα υπόλοιπα. Υπάρχουν και κάποιοι που ζουν προσωρινά σε μια χώρα, αλλά δεν ξέρουν αν είναι μια βεταβατική περίοδος ή αν ε, θα καταφέρουν να βρουν δουλειά και να μείνουν σε μια χώρα. Κοιτάξτε την αγορά εργασίας από χώρα σε χώρα, διαφέρουν. Στη Γερμανία είναι πιο εύκολο, σχετικά εύκολο να βρεις δουλειά, σε άλλα κράτη όχι. Έρχονται άνθρωποι στη Γερμανία, ψάχνουν δουλειά, δεν ξέρουν αν θα μείνουν τρει μήνες ή τη ζωή τους όλοι ε, και πώς ε, θα ξέρουν να ανοίξουν ένα λογαριασμό. Και πού είναι η εσωτερική αγορά και πού είναι η ευελιξία των ανθρώπων και η πρόσβαση ε, σε άλλες αγορές εργασίας και σε άλλα, άλλους τόπους για τη ζωή τους. Αυτό που με ενδιαφέρει επίσης είναι, όπως είπαν και κάποιοι προλαλήσαντες, να μην είναι μεμονωμένες οι τράπεζες που θα πρέπει να δίνουν αυτή την προσφορά ε, ε, ανακράτος μέλος για τον εξής απλό λόγο που ανέφερε η κυρία Λούλινγκ. Δεν θα πρέπει μια τράπεζα να τη ρετσινιά της τράπεζας των φτωχών ε, και ε, κάθε ε, τράπεζα μπορεί να εκπροσωπείται παντού ας πούμε στην Ήπεθρο είναι συγκεκριμένες σήμερα οι τράπεζες που έχουν υποκαταστήματα θα πρέπει να υπάρχουν όλες ε, οι τράπεζες να είναι υποχρεωμένες και αυτές που έχουν υποκαταστήματα παντού σε μία χώρα. Ένα τελευταίο, τα δύο, πολύ σύντομα, σε ό,τι αφορά τα τραπεζικά τέλη, θα πρέπει να υπάρχουν οροφές που θα ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές και μάλιστα διανόμου αυτό να κατοχυρώνεται και όχι μέσω του μηχανισμού των τραπεζικών τελών να αποκλείουν κάποιους ανεπιθύμητους πελάτες ή τράπεζες. Και τελικά αυτοί που απορρίπτονται από μια τράπεζα για το άνοιγμα ενός βασικού λογαριασμού θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κάπου να προσφεύγουν. Να τους αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι ε, ή ε, να ξέρουν για ποιο λόγο και τι ένομα μέσα έχουν στη διάθεσή τους για να προσφύγουν. Γιατί μόνο όταν ξέρεις γιατί σε απορρίπτουν μπορείς να διεκδικήσεις το δίκιο σου και να προσβάλλεις αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Uh, uh Jean-Paul Ευχαριστούμε Jean-Paul Merci, Madame la Quelques observations générales. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ μάλλον θα πάρω μια διαφορετική θέση από του υπόλοιπου, αλλά γιατί όχι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση στο δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το, για αυτό το κείμενο και για τους πολίτες. Το θέμα είναι να αποδείξουμε ότι απασχολούμαστε με τα ζητήματα που απασχολούν άμεσα την κοινωνία. Είχαμε συζητήσει κάποια από αυτά τα θέματα στο πλαίσιο της συζήτησης για την ε, υπηρεσία πληρωμών. Οι υπηρεσίες πληρωμών δεν είναι δημόσιο αγαθό, δεν είναι ε, δημόσια υπηρεσία, είναι μια ε, εμπορική δραστηριότητα, επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, απαιτήσει στους επιχειρηματίες της επιχειρήσης αυτού του κλάδου, οι οποίες να είναι υπερβολικές. Είναι λογικό να επιδιώκουμε την καταπολέμηση του ε, κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένου αυτού και μέσω της δημιουργίας ενός απλού βασικού λογαριασμού πληρωμών. Αλλά δεν θα πρέπει να αυξήσουμε το κόστος και τους περιοριστικούς όρους που επιβάλλονται σε, ε, στις τράπεζες ε, και κάτι που τελικά δεν θα έχει και αποτέλεσμα. Ας συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε το ΣΕΠΑ κόστισε περισσότερο ακόμα και από την ε, έναρξη κυκλοφορίας του ευρώ, του ευρώ. Σε επίπεδο ε, πληροφοριακών συστημάτων, σε επίπεδο ε, εκπαίδευσης του προσωπικού. Επομένως οποιαδήποτε καινοτομία ενδιαφέρουσα είναι, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το κόστος της. Και να σταθμίζουμε αυτό το κόστος σε σχέση με το όφελος που αποφέρει στην κοινωνία. Για να αποφασίζουμε τα Λόγω γνώσεως, εάν τελικά ε, υπάρχει λόγος, υπάρχει για παράδειγμα λόγος να να, να, προωθήσουμε αυτές τις ρυθμίσεις εάν ενδιαφέρεται μόνο ένας περιορισμένος μικρός αριθμός ε, καταναλωτών. Αναφερόμαστε στους φοιτητές, σε, μετανάστε τους εργάτες, σε όσους δεν γνωρίζουν αν θα ε, παραμείνουν ε, επαόριστον σε μια χώρα, αλλά μην υπεργενικεύουμε, δεν γνωρίζουμε τελικά πώ είναι οι καταναλωτές οι οποίοι θα ενδιαφέρονται να ανοίξουν τέτοιου τύπου λογαριασμούς. Επίσης να μην δημιουργήσουμε ένα υπερβολικά γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο τελικά θα κοστίσει. Και ποιος θα πληρώνει να λάβει αυτό το κόστος, ο ίδιος ο πελάτης της ε, τράπεζας. Χρειάζεται ε, τα ε, έγγραφα και ενημέρωση από την τράπεζα προς τον πελάτη να είναι ξεκάθαρη. Κάθε χρόνο μου στέλνει η τράπεζά μου έγγραφα ε, του γενικού όρου συναλλαγών, για να είμαι ειλικρινή, εγώ δεν του καταλαβαίνω. Εκεί μέσα υπάρχουν και όροι πολύ ε, ακατανόητοι. Δηλαδή, τελικά, όταν φτάνουμε από το ένα, το ένα άκρο είναι να μην έχουμε αρκετέ πληροφορίε, αλλά το άλλο άκρο είναι να φτάνουμε σε τελείω ε, τεράστια κατανόητα κείμενα. Άρα ας περιορίσουμε τη δράση μας σε αυτό που είναι ε, πραγματικά σημαντικό και σε αυτό που πραγματικά θα καταπολεμήσει τον κοινωνικό ε, αποκλεισμό και θα συμβάλλει σε μια ε, φυσιολογική ελεύθερη μετακίνηση προσώπων που θα ενθαρρύνει και την ελεύθερη αγορά. Φανταστείτε θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από όλα τα εστιατόρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν ένα μενού στι 28 γλώσσε, στι 24 συγγνώμη, επίσημες γλώσσες, μόνο και μόνο για να βοηθήσουμε την ε, κινητικότητα. Ε, φαντάζομαι πώ. όχι. Άρα παρόλο που έχει γίνει δημοφιλέ να κατηγορούμε τις τράπεζες, ε, είμαστε... Ε, ε, ας αυτοπεριοριστούμε, ας ζητήσουμε μόνο αυτά τα οποία είναι λογικό να ζητάμε. Συμφωνώ με αυτό που είπατε σε σχέση με τους γενικούς όρους συναλλαγών. Ε, τους, ε, ε, μάλιστα μια φορά είχα αποστείλει πίσω το σχετικό έγγραφο λέγοντας μάλλον θα αστείευεστε. Ε, πάρα πολύ γρήγορα. Ο κύριος Λάγκεν. Δεν είναι μόνο θέμα Βουλγαρίας-Ρουμανίας λέτε. Σε έξι κράτη-μέλη, τα εξή επτά, έχουμε νόμους ε, Γαλλία, κάτω χώρες, Δανία, ε, Σουηδία ε, και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. Δεν μπορείς με το ζόρι να τους αναγκάσεις. Είναι θέμα και νοοτροπίας, αλλά παραμένει κάτω ε, του 10% του πληθυσμού, ενώ στη Ρουμανία είναι 40% και στη Βουλγαρία 60% του πληθυσμού δεν ήθελα να το περιορίσω ή να κατονομάσω μόνο αυτές τις δύο χώρες, αλλά ακόμα και αν υπάρχουν ρυθμίσεις, ο κόσμος σου λέει δεν θέλω να ανοίξω λογαριασμό, τι να κάνουμε. Έχω κάνει αυτή την ε, πρόταση ε, κάθε τράπεζα να προσφέρει ένα τέτοιο λογαριασμό πληρωμών και δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις οι άνθρωποι. Παραδείγματα, στην Τουρκία επί σειρά ετών έγραφε στο διαβατήριο ε, υπήρχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για ορισμένες εθνικές ομάδες και ορισμένες θρησκείες και το έβλεπε ε, ο ελεγκτής στα σύνορα. Στο μεταξύ έχει αυτό ε, καταργηθεί και στη Γερμανία έχουμε ζήσει τέτοια ε, φαινόμενα. Άρχισε ε, με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και στη συνέχεια κατέληξε στην εξολόθρευση μιας ομάδας. Και στη Γερμανία ε, όποιος έπαιρνε επίδομα πρόενιας χωρίς να φαίνεται στο έμβασμα υπήρχε ένας έξτρα αριθμός και το ήξερε ο υπάλληλος της τράπεζας ότι είναι επίδομα που έρχεται από την πρόνοια αυτό το έμβασμα χωρίς να το καταλαβαίνει ο ενδιαφερόμενος. Ε, γι' αυτό ζητώ λοιπόν να αρθούν όλες οι διακρίσεις. Uh, το ήταν το σύντομο, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το φυλάδιο που μας έδειξες. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή της ΣΥΜΚΟ που έφτασε, στο μεταξύ στην εισηγήτρια. Το συζητήσαμε λίγο, αλλά έχετε κάνει και εσείς τροπολογίες ε, στην ε, Επιτροπή μας. Είπα ε, στην αρχή η αποσία σας ότι ανησυχούμε λίγο με το χρονοδιάγραμμα της ΙΜΚΟ. Αν δεν ψηφίσετε μέχρι τέλη του Νοεμβρίου, τότε μας χαλάτε τα σχέδια ε, να τελειώσουμε το θέμα αυτό εντός της παρούσης θητείας. Ε, δεν ξέρω αν μας βοηθάει αυτό. Αύριο συνεδριάζουν οι συντονιστές να το σημειώσουν παρακαλώ ε, οι πολιτικές ομάδες και να το ψηφίσετε στις 4 και 5 Νοεμβρίου. Δεν χρειάζεται να περιμένετε την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων για να αρχίσετε. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Θα πάει στην επόμενη θητεία και είναι κρίμα. Θα έχουμε αποτύχει εμείς. Κύριε Γκέπχαρτ, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, λυπάμαι πραγματικά πολύ που η διάσκεψη των Προέδρων εργάζεται με τέτοιους βραδείς ρυθμούς και παίρνει τέτοιες αποφάσεις μετά από τόσο καιρό. Και σε δική μας επιτροπή αρχίζουμε τις εργασίες μας ε, όταν λαμβάνουμε επισήμως την άδεια να το κάνουμε. Εγώ προσπάθησα να το αλλάξω αλλά δεν γίνεται. Η πλειοψηφία των συντονιστών το βλέπει διαφορετικά και δυστυχώς έχουμε περιέλθει στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Η, μετάφραση συγγνώμη, της έκθεσής μου θα έρθει μόνο στις 4 Νοεμβρίου, μια στιγμή να δω ακριβώς τις ημερομηνίες και γι' αυτό δεν μπορούμε να ψηφίσουμε στις 5 δεν γίνεται, δεν προλαβαίνουμε, δεν χωράει, γιατί οι συνάδελφοι στην Επιτροπή μας είναι ε, και στο άρθρο 50 συνεργασία των Επιτροπών και δεν μπορώ να απαιτήσω από τους συναδέλφους να μην κάνουν και τροπολογίες. Δεν γίνεται, απλούστατα δεν προλαβαίνουμε. Να σας βοηθήσω όσο μπορώ και για να το κάνω αυτό έδωσα την έκθεσή μου στα αγγλικά παρακαλώ. Ε, αλλά αύριο στην ε, Επιτροπή μας, στη συνεδρία των συντονιστών συγκεκριμένα, θα το συζητήσουμε, αλλά φοβούμαι ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε πριν τις 28 Νοεμβρίου στην ΙΜΚΟ. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά τι να σας κάνω. Δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα αυτό, αλλά στη διαδικασία που έχουμε γενικά στο κοινοβόλιο. Πώς να το πω. Η διάσκεψη των Προέδρων τα ορίζει αυτά τα θέματα. Ε, επί της ουσίας τώρα και από ε, τη Σκοπιά ΙΜΚΟ που είναι και εσωτερική αγορά αλλά και προστασία των καταναλωτών και οι δύο πολύ σημαντικοί τομεί για μας. Εγώ έθεσα βεβαίω ιδιαίτερα το κέντρο βάρους στο εξή να έχουμε ε, εσωτερική αγορά όχι μόνο για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη αλλά και για τους πολίτες και θα πρέπει να υποφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς οι πολίτες μας και ως κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση και να φροντίσουμε κι εμείς να υπάρχει δυνατότητα διασυνοριακής αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού και μάλιστα όσο γίνεται πιο εύκολα. Η μεταφορά δηλαδή από το ένα κράτος στο άλλο, ε, όπως είναι εξίσου εύκολο και εντός του ιδίου κράτους. Κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που είπε ο Πέτερ Ζήμων. Συμφωνώ πολύτος. Πρόκειται για μια σειρά πάρα πολύ διαφορετικών περιπτώσεων. Υπάρχουν ε, άστεγοι που δεν έχουν διεύθυνση και γι' αυτό αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Παρόλο που θέλουν πολλές φορές. Επίσης υπάρχουν κάποιοι πολίτες σε Ρουμανία και Βουλγαρία που συχνά δεν έχουν την ευκαιρία καν διότι στην Ήπεθρο δεν υπάρχουν τράπεζες. Ε, ε, ε. Πού να πας να ανοίξεις αν δεν έχει υποκατάστημα όταν ζουν συνήπεθρο οι άνθρωποι. Βέβαια τώρα έχουμε νέα μέσα επικοινωνίας που το επιτρέπουν. Στα πλαίσια των 20 ετών της εσωτερικής αγοράς που γιορτάσαμε πέρυσι, βλέπουμε και φοιτητές Εράσμου που λέγουν ότι θέλουν να υπογράψουν ένα μισθωτήριο συμβόλαιο και σου λέει δεν γίνεται πού είναι ο τραπεζικός σου λογαριασμός. Και πάνε στην τράπεζα και λέει η τράπεζα «Α, μα δεν έχεις διεύθυνση, πώς θα σου ανοίξω λογαριασμό». Και ε, οι άνθρωποι που ε, κυκλοφορούν οι φοιτητέ με τον αίρεσμο, δεν μπορούν να έχουν τέτοια αντιμετώπιση. Είναι ολέθριο αυτό για την εικόνα, το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πραγματικά δεν πρέπει να έχουμε διακρίσεις εκεί. Και κάτι ακόμα. Ε, επίσης, πραγματικά στην ουσία να μην γίνονται διακρίσεις. Δηλαδή, όχι κάποιες μεμονωμένες τράπεζες να προσφέρουν αυτό, αλλά όλες ε, οι τράπεζες που παρέχουν ε, υπηρεσίες λιανικής ε, σε ιδιώτες, τις άλλες τις επαγγελματικές αφήνω στην άκρη. Αλλά όσε δίνουν τέτοια δυνατότητα σε ιδιώτες θα πρέπει όλες να προσφέρουν ε, το λογαριασμό αυτό, ακριβώς για να μην υπάρχει καμία διάκριση και μεταξύ των τραπεζών. Γιατί τέτοιου βασικούς λογαριασμούς πληρωμών θέλουμε να τους προσφέρουν όσο γίνονται φτηνότερα, για να μην πω και δωρεάν, στο βαθμό που επιτρέπεται και γίνεται αυτό, γιατί ο φτωχό κόσμο να έχει μια δυνατότητα να ανοίγει λογαριασμό. Ένα τελευταίο, γιατί βλέπω ότι δεν έχετε και πάρα πολύ χρόνο, είναι η ενημέρωση και βέβαια είναι απαραίτητη η πληροφόρηση έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες τι τους περιμένει όταν ανοίγουν ένα τέτοιο τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά μόνο μερικά από τα σημεία που είχα να σας παρουσιάσω και στις τροπολογίες μου έχω καταθέσει και προσπάθησα πραγματικά να εργαστώ πάρα πολύ γρήγορα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, αλλά θαύματα δεν κάνω. Και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Um, λοιπόν, για το χρονοδιάγραμμα είπατε στις Τέσσερις με πέντε θα είναι έτοιμη μεταφρασμένη έκθεση ή τροπολογίες. Ε, για τις τροπολογίες πότε είναι η προθεσμία. Την έκθεση μου την έχω δώσει. Δυστυχώς για τις μεταφράσεις στο Κοινοβούλιο έχουν επιμηκυνθεί η ε, περίοδοι μετάφρασης γιατί κάνουμε οικονομίες και περικοπές και για τις τροπολογίες στις 4 Νοεμβρίου ε, θα έχουμε στην ΙΜΚΟ τη μετάφραση, παρόλο που εγώ έχω ήδη δώσει την έκθεσή μου. δεν το καταλαβαίνω. Και πότε είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών? Εβελίν, πότε, πότε λίγη η προθεσμία? Ε, λοιπόν, να το ξαναπώ από την αρχή. Πάμε πάλι. Έχω δώσει το κείμενό μου στις 14 Οκτωβρίου ε, το σχέδιο γνωμοδότησης συζητείται. 16 Οκτωβρίου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 4 ε, Νοεμβρίου ε, θα έχουμε τις μεταφράσεις και στις 5 Νοεμβρίου θα το συζητήσουμε και στις 28 Νοεμβρίου είναι η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Γιατί από τις 4 μέχρι τις 28 δεν θα υπήρχε άλλη συνεδρίαση. Τη συγκόλιο θα έλεγα να συζητηθεί το δικό μου θέμα και να ψηφιστεί, αλλά δεν γίνεται. Uh, Ωραία, άρα η τροπολογία σας θα είναι έτοιμες και μεταφρασμένες στις 4 και τις 5. Όχι, όχι. Όλες, όλες. Ναι, σωστά. Δηλαδή αυτό είναι πριν την ψηφοφορία στη δικιά μας επιτροπή και ως... Ε, αρμόδια επιτροπή θα έχουμε την τελική ψηφοφορία και θα έχουμε στη διάθεσή μας και τις δικές σας τροπολογίες. Αυτό λοιπόν προτείνω να έχουμε ένα ε, ολοκληρωμένο κείμενο όταν εμείς θα ψηφίσουμε για να μην ε, ε, δημιουργηθεί πρόβλημα αν εσεί έχετε ψηφίσει κάτι διαφορετικό θα το λάβουμε υπόψη μα στο τριμερή διάλογο και αν παραμείνουν κάποιε διαφωνίε, θα μπορούσαμε να τι λύσουμε στην Ολομέλεια. Έτσι το βλέπω κάπως να το λύνουμε το θέμα. Εκτό βέβαια εάν βρούμε έναν τρόπο να συμπεριλάβουμε τι τροπολογίε τη δικέ σα στο δικό μα κείμενο. Με συμβιβαστικέ τροπολογίε, για παράδειγμα. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ειδική ε, συνάντηση στο Στρασβούργο είναι κάτι που το έχει κάνει στο παρελθόν η Επιτροπή Οικονομικών για να ε, υποχρεώσει άλλες επιτροπές να κινηθούν πιο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Γιούργεν Κρούτε, που είναι εισηγητής μας αυτή τη στιγμή της ημέρας μάλλον του ηλιοβασιλέματος, θα σας δώσω το λόγο για να ολοκληρώσετε την συζήτηση. Δεν θα μπω τώρα στα θέματα του αριστερού φιλελευθερισμού, θα το συζητήσουμε άλλη ώρα. Ήθελα να κάνω μια διαπίστωση πρώτα και να ευχαριστήσω βέβαια για τα όσα είπατε. Είναι επικοδομητικά όλα αυτά. Κανείς δεν εκφράστηκε κατά ε, της ε, πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η βασική διαφορά είναι πώς θα έχουμε μια ισορροπία λογική ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ε, προσπάθεια, το ευρωπαϊκό πλαίσιο και την επικουρικότητα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Δεν το βρίσκω και ανυπέρβλητο εμπόδιο για να σας πω την αλήθεια. Ε, για τη γραφειοκρατία συμφωνώ, πραγματικά να μην το βαρύνουμε πάρα πολύ, παρόλα αυτά όμως πρέπει να πω ότι να προσέξουμε για την πρόσβαση. Δηλαδή, να μην είναι και αυτό υπερβολικά γραφειοκρατικό. Για την πρόσβαση υπάρχουν πολλές προτάσεις και πολλές ιδέες και πολλές ρυθμίσεις που, πώς να το πω, μάλλον είναι φιλικές και προς τη γραφειοκρατία και παραεχθρικές. Και καλό θα ήταν και εδώ να έχουμε κάποιο μέτρο. Να πω κάτι που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι για τις 28 χώρες. Εγώ δεν θέλω να γίνω διάσημος από αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι ένας Βρετανός gentleman σε κάποια λέσχη μπορεί να βάλει στοίχημα με τους φίλους του εκεί ότι θα ανοίξει λογαριασμό σε 28 χώρες. Το θέμα είναι το εξή. Ένας φοιτητής, ένας εργαζόμενος που αλλάζει χώρα είναι από μια άλλη χώρα και πάει σε μια γειτονική για περιορισμένο χρόνο και χρειάζεται τραπεζικό λογαριασμό. Δεν μπορούμε να πούμε μα αυτός έχει λογαριασμό σε άλλη χώρα. Άρα δεν μπορεί να ανοίξει καινούριο εκεί που σπουδάζει ή εργάζεται, βασικό λογαριασμό, αλλά εκεί μπορεί να το χρειάζεται. Ε, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Γιατί έτσι δημιουργούνται και οι δεσμοί με τη χώρα. Πώς θα αποδείξεις το δεσμό με τη χώρα ε, εκ των προτέρων δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί η δυνατότητα αν κάποιο θέλει να πάει σε άλλη χώρα. Αλλά στη χώρα του να μην κλείσει το λογαριασμό του, γιατί εκεί είναι η οικογένειά του, οι δεσμοί και το σπίτι του, να μπορεί να ανοίγει και ένα δεύτερο λογαριασμό. Γιατί έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που θέλουμε να λύσουμε. Αλλά να μην λέμε ότι αν έχει κάπου ένα λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην έχει πουθενά άλλου. Δεν λειτουργεί αυτό. Ή όπως λέει η Λούλινγκ, να μπορείς να έχεις βασικό λογαριασμό μόνο στην πατρίδα σου. Μα τότε καταστρέφεις αυτή την ιδέα. Κάποιος που ζει σε μια γειτονική χώρα για περιορισμένο χρόνο να μην ανοίγει τέτοιο λογαριασμό, τότε καταστρέφεται η ίδια ιδέα. Δεν ξέρω κάπως αλλιώς να το διατυπώσουμε. Ειλικρινά δεν βλέπω, επαναλαμβάνω, κανένα ε, τεράστιο εμπόδιο που να μας αποτρέπει από το να συμφωνήσουμε. Και ένα τελευταίο. Στο Στρασβούργο συναντηθήκαμε με την Όλμπικ, μας κάλεσε ο Ζάνρο. Η κυρία Ισαΐα από τη Φιλανδία είπε ότι στο μεταξύ στη Φιλανδία ε, ε, μισθοί ε, και χρήματα και συντάξεις πληρώνονται μόνο με τραπεζικό λογαριασμό. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Το είχα πει και στην πρώτη τοποθέτηση ότι στην Ιταλία από 1000 ευρώ και πάνω όλοι οι λογαριασμοί θα πρέπει να γίνονται τραπεζικά όλες οι πληρωμές για να ελέγχετε το μαύρο χρήμα, το ξέπλυμα κτλ. Ό,τι έχεις να πληρώσει πάνω από 1000 ευρώ ο τραπέζης. Όλο και περισσότερο ε, απαιτούνται να έχεις ένα λογαριασμό, άρα θα πρέπει ο πολίτης να έχει το δικαίωμα να ανοίγει λογαριασμό. Αυτά είναι αλληλένδετα, πιστεύω. Και δεν είναι μόνο ένα θέμα κοινωνικής πολιτικής που είναι και αυτό, ε, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής πολιτικής, αλλά όλο και περισσότερη γίνεται ηλεκτρονική πληρωμή μέσω ε, ε, τραπεζικού λογαριασμού και όχι σε μετρητά. Και για τις χώρες που ανέφερε ο Λάγκεν, Ρουμανία και Βουλγαρία, από ό,τι φαίνεται ο κόσμος εκεί δεν εμπιστεύεται το τραπεζικό σύστημα, γι' αυτό δεν ανοίγει λογαριασμό. Αλλά αν ζούμε σε μια εσωτερική νέα αγορά, θα πρέπει και τον τραπεζικό τομέα και το χρηματοπιστωτικό πάνω κάτω να τον ε, ομοιογενειοποιήσουμε και να έχουν ε, όλοι εμπιστοσύνη στις τράπεζες, αλλιώς καήκαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ε, μια κάπως ε, στοιχειοδός εναρμονισμένη εσωτερική αγορά και λειτουργούσα. Αυτά τα άλλα διαφάνεια και τα λοιπά είναι πολύ σημαντικά για την εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση και αυτό ήθελα να προσθέσω. Α, ένα τελευταίο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πατρίδα μου, σε μια γειτονική πόλη στη δικιά μου, εν πάση περιπτώσει, συζήτησα με κάποιους αστέγους και ε, έκανα μια βόλτα στην πόλη και μου είπανε ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι από την Ανατολική Ευρώπη που έρχονται στη Γερμανία και για πολύ καιρό δεν έχουν ε, ε, σπίτι και στεγάζονται ε, σε ιδρύματα που είναι για στέγους, αλλά εργάζονται. Αλλά επειδή δεν ξέρουν πόσο θα μείνουν, πόσο θα δουλέψουν, δεν έχουν ψάξει για σπίτι, δεν έχουν βρει σπίτι, αλλά χρειάζονται πηγόντως τραπεζικό λογαριασμό. Δεν είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής, ε, ούτε είναι μειονεκτική ομάδα, είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν ε, αλλά δεν έχουν μόνιμη κατοικία στη Γερμανία ή κάπου. Και σε ό,τι αφορά την κατοικία θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην αποκλείουμε τέτοιους ανθρώπους με λάθος ε, διατύπωση. Αυτά. Και νομίζω ότι Τέλειωσα ακριβώς στις 6.30 ώρα ε, και σταματώ εδώ και θα τα ξαναπούμε άλλωστε με τους σκιοδησίγητες. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Earlier in the... Πολύ σας ευχαριστούμε. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα τελειώσουμε πολύ νωρίτερα από τις 6, αλλά μας διασκέδασε τόσο πολύ η τελευταία έκθεση που φτάσαμε στις 6.30. Θα ψηφίσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα γίνεται. Είχαμε και εναλλακτικέ ημερομηνίε, 14 Οκτωβρίου ήταν αρχικά, αλλά ούτε καν ε, τι τροπολογίε σου και τι συμβαστικέ θα έχουμε τελειώσει τότε. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσο εσείς εργάζεστε για να καταλήξετε συμβαστικές τροπολογίες, ε, θα δούμε και εμείς αν προκύψει κάτι καινούργιο, θα σας στείλουμε το χρονοδιάγραμμα αν μπορείτε να πιέσετε τους συναδέλφους στη ΣΥΜΚΟ, κάντε το. Ευχαριστούμε. Κάποια στιγμή στο μέλλον, λέει η Πρόεδρος, θα ξανασυνεδριάσουμε. Δεν βλέπω τώρα. 30 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα, Δευτέρα. Ευχαριστώ.